Good morning, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Παρακαλώ να καθίσετε. Για να ξεκινήσει αυτή η πολύ σημαντική συνεδρίαση. We expect more... Περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα να εμφανιστούν και άλλα μέλη και από τις δύο επιτροπές, αλλά ας μην ε, χασομεράμε και ας αρχίσουμε. Αγαπητέ κύριε Όσβαλτ, Επίτροπε Κρέτσου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τιμή μου που σας ε, καλωσορίζω στην Κοινή Επιτροπή Reggie Cotter που έχει θεσμοθετηθεί ως ετήσιος χώρος συζήτησης μεταξύ των μελών της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών στη διάρκεια της θητείας μας. Αν η μελέτη του νέου πακέτου των προτάσεων μας οδηγεί στο να συζητήσουμε το νέο αυτό κείμενο με την Επίτροπο Κρέτσου. Θεωρώ ότι η σημερινή συνεδρίαση θα αποτελέσει ευκαιρία για παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα περισσότερο παραποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας, της δημογραφικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, θεμάτων ασφαλείας, την κρίση της μετανάστευσης και του προσφυγικού, την, το Brexit και τη γεωπολιτική αστάθεια. Οι αξίες και οι ανθρωπιστικές αρχές επί των οποίων ε, στηρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζονται. Οπότε είναι μεγάλο απίτευμα το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής παραμένει ένα από τα βασικά μέσα που έχει έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι περιφέρειες και οι πόλεις για να προωθήσουν την ισχυρή και βιώσιμη οικονομία στην Ευρώπη για τη μυρία νέων θέσεων εργασίας, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή εξάρτηση, όπως επίσης και θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Γιατί οι αρχές αυτές προέρχονται από, το γεγονός ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την εθνική ανάπτυξη καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες διαφόρων περιοχών και περιφερειών και να τα φέρουμε στους πολίτες. Η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή, αποτελεί καλή βάση συντονισμού και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Δυστυχώς ε, τα, οι περικοπές έχουν ε, γίνει κυρίως στην ε, πολιτική συνοχής και την αγροτική πολιτική. Στο, αυτό το πλαίσιο, το οποίο εγκρίθηκε το Μάιο του 2018, έχει οδηγήσει το Κοινοβούλιο να επαναλάβει την πρότασή του για επιπλέον χρηματοδότηση βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν διάφορες πολιτικές όπως επίσης και η διατήρηση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής τουλάχιστον στο επίπεδο της περίοδου 2014-2018. Μία από τις βασικές αρχές της νομοθετικής πρότασης της περίοδου 2021-2027 θα είναι να ενισχυθούν οι συμπληρωματικότητες των ταμείων όπως προτείνεται από τον νέο κανονισμό κοινών διατάξεων και άλλες διατάξεις θα ήθελα να προτείνω η πρόταση για την εξυγχρονισμένη και αναθεωρημένη πολιτική συνοχής στοχεύει στην βελτίωση της στόχευσης και τη συγκέντρωση της πολιτικής αυτής σε συγκεκριμένους στόχους. Ο, προτε... ο οδηγός με τους ενιαίους κανόνες ε, που περιλαμβάνει και, περιλαμβάνει και τα άλλα ταμεία και τα χρηματοδοτικά μέσα και συνάδει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πολιτική συνοχής του 2020 και την 7η έκθεση συνοχής. Ενισχυμένη σχέση μεταξύ των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομικής διακυβέρνησης θα βοηθήσουν την υλοποίηση των ταμείων. Οι τοπικές, αστικές και ε, εδαφικές αρχές θα υποφεληθούν περισσότερο μέσω των στρατηγικών που θα αναπτυχθούν επί τόπου. Αντιμετωπίζουμε τις επερχόμενες ε, ευρωπαϊκές εκλογές και επικεντρωνόμαστε στην ε, μελέτη νομοθετικών προτάσεων ώστε να δώσουν αυτές ε, στην Ευρώπη και τους πολίτες της μια καλή προοπτική για το μέλλον. Η Επιτροπή μας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια σειρά από νομοθετικά θέματα. Στο σκοπός μας είναι στην Επιτροπή να ψηφιστούν όλα τα νομοθετικά θέματα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων η Επιτροπή των Περιφερειών καλείται να παραβρεθεί στη συνεδρία της Επιτροπής μας και να παρουσιάσει τις γνωμοδοτήσεις κατά τη διάρκεια της σύνταξης των εκθέσεων που αφορούν το πακέτο συνοχής. Υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου στο διάστημα αυτό στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να παραδώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τη γνωμοδότησή μας. Ελπίζουμε ότι μετά τις εκλογές το νέο Κοινοβούλιο θα συνεχίσει με, την, με τον ίδιο ρυθμό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να παρουσιάσει στους Ευρωπαίους πολίτες ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πακέτο που θα είναι οριστικοποιημένο και που θα επιτρέψει να ξεκινήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση νέα προγραμματική περίοδος. Ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι παραγωγική. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Όσβαλτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μιχαήλοβα. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Είχα ετοιμάσει μια ομιλία αλλά είπατε τα περισσότερα. Να προσθέσω όμως κάτι από πλευράς Επιτροπής Περιφυρών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την παραδοσιακή συνάντηση εδώ και κάποια χρόνια μεταξύ της Κότερ και της Ρέτζι. Είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό που είναι παρούσα και η κυρία Επίτροπος για να συζητήσει μαζί μας. Γιατί εδώ και χρόνια αγωνιζόμεθα για τη συνοχή δεν ήταν ε, επαρκώς παρούσα στις προτάσεις Γιούνκερ και γι' αυτό δημιουργήσαμε τη Συμμαχία για τη Συνοχή ούτως ώστε και η κοινή γνώμη και η Επιτροπή και όλοι να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η συνοχή για όλους τους συμπολίτε μας και ιδιαίτερα τώρα που επίκυνται οι ευρωεκλογέ. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν γιατί αλλιώ δεν θα προκύψει ένα σωστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συνοχή θα μπορούσε να οθήσει τους πολίτες να ψηφίσουν γιατί αποδεικνύει αυτό το οποίο πάντα προωθούμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία άρα έχει σημασία να το καταλάβουν και οι ψηφοφόροι Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτούς τους κανονισμούς Υπάρχουν εισηγητέ και από τις δύο πλευρές για τις προτάσεις τη Επιτροπής. Οπότε, στόχος μας είναι μέσω της συνεργασίας μας να προκύψει ο βέλτιστος ε, κανονισμός για την Ευρώπη και για τους τελικούς δικαιούχους για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας ότι τους βοηθάνε αυτή η προσπάθεια. και χαίρομαι που η πολιτική συνοχή αφορά όλες τις ε, περιφέρειες. Βεβαίω υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι απλώς ο κανονισμός. Είναι να επιδιώξει και να επιτύχει την απλούστευση για την οποία ε, έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες. Άρα δεν είναι το θέμα μόνο του κανονισμού, αλλά και των κατευθυντηρίων γραμμών, γιατί είναι περίπλοκη η κατάσταση. Ο στόχος μας είναι να προωθηθούν τα προγράμματα που θα βοηθήσουν καλύτερα, που είναι πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε περιοχής. Χρειαζόμαστε μια ευελιξία και μια ενοποιημένη προσέγγιση. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια εδαφική προσέγγιση. Λοιπόν, να μην πω περισσότερα. Έχουμε τους εισηγητές μας και τα δύο όργανα. Αναβάλαμε για ένα μήνα ε, την συνεδρίαση της Επιτροπής μας ΚΟΤΕΡ για να διεξαχθεί μετά από τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ούτως ώστε να συζητήσουμε πιο εμπεριστατωμένα στη δική μας συνεδρίαση κατόπιν. Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Όστβαλντ. Θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο, κυρία Κρέτσου. Με πολύ προσμονή θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας, ε, γιατί χαιρετίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάντα μας ενδιαφέρει να το συζητήσουμε. Μα και εμένα είναι χαρά μου Ευχαριστώ και την ε, κυρία Μιχαήλοβα και τον κύριο Όσφαλτ, αξιότιμα μέλη και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφέρειων. Όπως είπα, είναι πάντα χαρά μου να συζητώ με εσά. Δεν είναι η συνήθις κατάσταση όμως τώρα. Συνεδριάζουμε μόλις υποβλήθηκε η πρότασή μας για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πρέσιο για την περίοδο 21-27. Την έχετε λάβει. Όπω και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι δύο συνομοθέτες. Η στήριξή σας είναι, όπως και στο παρελθόν, ουσιώδης. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή. Και εκτιμώ ιδιαίτερα τον ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο συζητάτε το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ο κύριος Όσβαλντ μας ε, θύμισε τη συμμαχία για τη συνοχή. Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Η ισχύ εν ενώση και μέσω αυτής της ε, ισχύω στείλαμε ένα μήνυμα προς όλους τους ε, ενδιαφερομένους φορείς. Και πρέπει να συνεχίσουμε και στο μέλλον με την ίδια αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι επιτύχαμε να είναι η κύρια επενδυτική προσπάθεια συνοχή της Ένωσης. 373 δις προβλέπονται. Θα είναι βασικός ε, παράγων για τον εξυγχρονισμό της Ένωσης και δεν είναι μόνο απλώς πιστώσεις. Είναι έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, των αξιών και της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε πολλούς, ε, πολλά ορόσημα στην ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και πιστεύω ότι και αυτό θα είναι άλλο ένα ορόσημο στο δρόμο για τον εξυγχρονισμό. Όπως ξέρετε, η πολιτική αυτή ξεκίνησε το 1975. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, αν θυμάμαι καλά. Άρα χρειάζεται προσαρμογή. Ευχαριστώ πολύ για την ε, στήριξή σας και σας παρακαλώ να συνεχιστεί αυτή η στήριξη σε αυτή την προσπάθεια αναβάθμισης. Όπως είπατε πρέπει να είναι πιο φιλικές προς το χρήστη οι προτεραιότητες και θεματική εστίαση στις βασικές προκλήσεις και φυσικά απλούστευση, περισσότερος δυναμισμός, ούτως ώστε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Το εχειρίδιό μας για τις προτεραιότητες είναι τώρα πιο αποτελεσματικό όπως όλοι ξέρουμε ακόμη και μια απλή συσκευή όπως τα smartphone ε, μπορεί να είναι πιο, πολύ περίπλοκα για τον χρήστη. Έχουμε πέντε λοιπόν τώρα απλές προτεραιότητες που θα τις εκφράσω με μια πολύ ωραία πρόταση. Μια ευφυή, πράσινη, χαμηλού άνθρακα, κοινωνική και συνδεδεμένη Ευρώπη που να είναι κοντά στους πολίτες. Α, αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν κάνουμε τεχνητούς διαχωρισμούς πλέον για τις προτεραιότητες του στόχου 1 όπου έχουμε την καινοτομία, την ε, ψηφιοποίηση, τις δεξιότητες, τις μικρομεσαίες, την εκπαίδευση και την δυνατότητα αποτελεσματικότητας. Στο παρελθόν θα ήταν χωριστές προτεραιότητες. Αυτό τώρα το, ο νέος μας κατάλογος είναι πιο εύκολο και να ε, αξιοποιηθεί για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Γιατί κάνουμε πολλά, αλλά δεν ενημερώνουμε ε, πολλές, φορέ φορές σωστά τους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Γιατί είναι κρίμα όταν βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο 70% των πολιτών της Ένωσης όταν πηγαίνουν σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποιο σχολείο, όταν οδηγούν σε κάποιο δρόμο, δεν ξέρουν ότι έχουν ε, οικοδομηθεί με ευρωπαϊκή συμβολή. Πέντε λοιπόν απλέ προτεραιότητες. Πέντε καλύτερε από έντεκα. Πιο εύκολο να γίνουν κατανοητέ, ε, πιο εύκολο για την ενημέρωση, πιο εύκολο για να συμπεριληφθούν στι διάφορες πλατφόρμες. Βεβαίως, πέρα από το ότι είναι φιλικές οι δράσει μα προς το χρήστη, έχουν αλλάξει και, έχει αλλάξει και η Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ευφιέστερη Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργηθούν τα θεμέλια για αυτήν την ευφιέστερη Ευρώπη. Ποιες είναι οι εταιρείε στην πρωτοπορία σήμερα στον κόσμο. Είναι διάφοροι γίγαντες που όμως έχουν πολύ σύντομη ιστορία. Ιδρύθηκαν πριν από μερικά χρόνια. Πολλές φορές στον καράζ ενός ανθρώπου. Εκεί έπεσε ο δημιουργικός σπόρος σε γόνιμο έδαφος μέσω ε, της δυνατότητας χρηματοδότησης ε, που βεβαίως βασίζεται και σε μια περιφερειακή συγκέντρωση πρωτοβουλειών. Θέλουμε λοιπόν στις περιοχές μας, στις περιφέρειές μας να υπάρχουν αυτοί οι επιχειρηματίες που είναι ο αναγκαίος σπόρος για την αυριανή οικονομία. Και θα βοηθήσουμε ούτως ώστε να προκύψει το μόνιμο έδαφος για αυτούς ε, τους σπόρους μέσω της χρηματοδότηση για την έναρξη εταιριών, τη στήριξη στις, για την είσοδο στι αγορές για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε έναν όλο και πιο τεχνολογικό κόσμο. Δύο προκλήσεις έχουμε για να μετατραπεί, να μεταμορφωθεί η οικονομία στις περιφέρειές μας. Το ένα το ανέφερα, είναι η τεχνολογική, ε, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός αλλά επίση πρέπει να περάσουμε και στην οικονομία χαμηλού άνθρακα. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο πράσινη, χαμηλού άνθρακα. Δηλαδή περισσότερη ενεργειακή απόδοση και περισσότερη χρήση ανανεωσίμων. Πιο ευφυή ενεργειακά συστήματα. Και είμαι πεπισμένη ότι η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί του κόσμου σε αυτές τις τεχνολογίες. Τρίτον, απλούστερη και πιο δυναμική εφαρμογή των ε, νομοθεσιών μας. Πρέπει να έχουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό λοιπόν, σύστημα εφαρμογής. Κάτι που θα ακούσετε πολλές φορές, θα αναφερθώ πολλές φορές στα smartphone. Τι κάνουμε με ένα smartphone. Αν δεν έχουμε wifi τι κάνουμε. Αν είναι αργή η σύνδεση τι κάνουμε. Όχι. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει χρόνος αναμονής. Πρέπει να λειτουργούν οι τεχνολογίες μας. Πρέπει να εξαγάγουμε διδάγματα από το παρελθόν για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Και σας είμαι ευγνώμων, γιατί μας στηρίξατε όταν είπα ότι πρέπει να υπάρξει ριζική απλούστευση. Και κάναμε πολλή δουλειά μαζί σας για να μειώσουμε την γραφειοκρατία Είχαμε αυτή την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλούστευση και προτείνουμε ένα πολύ πιο φιλόδοξο και ορθολογικό πλαίσιο. Θέλουμε ε, η εστίαση να είναι όχι στις διαδικασίες αλλά στα αποτελέσματα. Έτσι βοηθάμε τους δικαιούχους να ασχοληθούν κυρίως με την εφαρμογή και όχι με την ε, συμπλήρωση εντύπων. Δεν είναι δυνατόν κυρίως να ασχολούνται με τις διαδικασίες, την υποβολή εκθέσεων και, τους, και τα τιμολόγια αυτοί που κάνουν τη δουλειά, αυτοί που εφαρμόζουν τα προγράμματα. Θέλουμε να εστιάζουμε στα αποτελέσματα, με δημιουργικότητα. Κάποια άλλη βασική κατευθυντήρια αρχή, πολύ σημαντική σήμερα, σε αυτή την ε, περίοδο που ενέχει τόσες προκλήσεις και αναστατώσεις. Το πιο σημαντικό είναι εμπιστοσύνη. Με βάση την εμπειρία τον μάνατζερ πρέπει να τους ε, σεβόμεθα δεν πρέπει να είμαστε αλαζονικοί να θεωρούμε ότι εμείς εδώ στις Βρυξέλλες ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τους δίνουμε πολύ περισσότερο περιθώριο να προσαρμόζουν τα προγράμματα στις ανάγκες τους. Πρέπει να σεβαστούμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στις τοπικές αρχές οι οποίες ε, έχουν καλύτερη γνώση ακόμη και των χείριστων συνθήκων. Οι προτάσεις μας για την απλούστευση είναι ευρείες και μακρόπνοες. Δεν έχω χρόνο να τις αναφέρω όλες. Αλλά υπάρχει ένα χειρίδιο για την απλούστευση που περιέχει 80 βασικά μέτρα απλούστευσης. Σας ευχαριστώ για την θετική αντίδραση από πλευρά σας. Με πολύ χαρά συζήτησα με πολλά ε, από τα μέλη και των δύο οργάνων και με πολλούς άλλους ενδιαφερομένους φορείς και ακούω πολύ στήριξη για την ε, προσπάθεια απλούστευσής μας και θα βασιστώ ιδιαίτερα και τους επόμενους μήνες στη στήριξή σας όταν θα συζητηθούν οι κανονισμοί αυτοί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Χρειάζομαι, πραγματικά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ξέρω πολύ καλά ότι και τα δύο όργανα πιέζουν για να υπάρξει ταχεία συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογέ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει και το Συμβούλιο. Πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν. Είναι ζωτική σημασία να υπάρξει συμφωνία για το ΠΔΠ πριν τι ευρωεκλογέ. Όχι λόγω των ευρωεκλογών, αλλά γιατί αλλιώ θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Γιατί υπάρχει κίνδυνος εάν δεν αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2021 το νέο ΠΔΠ θα πρέπει να υπάρξει εθνική χρηματοδότηση 100% των κάποιων προγραμμάτων. Άρα πρέπει να υπάρξει συμφωνία κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας. Όπως ξέρετε, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δύο εξωτερικούς παράγοντες επίσης. Αλλά ο πρώτος είναι ότι καθυστέρησε η, εφαρμογή, η έγκριση της νομοθεσίας την 1η Δεκεμβρίου του 2014 και μετά δεν είχαμε επαρκή χρόνο γιατί έπρεπε να υπογραφούν ε, και οι συμφωνίες εταιρική συνεργασίας και να γίνουν σεβαστές και οι Οπότε μας έμεινε μόνο ένας χρόνος. Δεν κρύβομαι. Σας το λέω ανοιχτά. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Ε, η αλλαγή πάντα κοστίζει. Και γι' αυτό πολλοί προσπαθούν ορισμένες φορές να μην αλλάζουν, να μην αγοράσουν το νέο πιο σύγχρονο κινητό που μπορεί να τους βολεύει αλλά δεν έχει μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να με βοηθήσετε υπενθυμίζοντας και εσείς ε, στα κράτη-μέλη ιδίω ότι το να μείνουμε στο παλιό θα έχει μεγάλο κόστος. Πρέπει λοιπόν το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και η νέα νομοθεσία να ισχύσουν τάχιστα για να υπάρξει περισσότερη απλούστευση και ευελιξία. Και είμαι πολύ περήφανη για όσα επιτύχαμε. Πριν από ένα-δύο χρόνια, όταν τα συζητούσαμε, εδώ σε αυτό το πλαίσιο, συζητούσαμε τι θα γίνει με το Brexit. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, ο δεύτερο καθαρό ε, συνεισφορέα. Ε, και αναρωτιόμαστε γιατί θα κάναμε για την ασφάλεια στα σύνορά μα. Γιατί για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβαινε σε αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε την ευρύτερη χρηματοδότηση για τη συνοχή, 373 δις όπως είπα, που, καλύπτει, που καλύπτουν όλες τις περιοχές και αυτό είναι σημαντικό γιατί το συζητήσαμε και αυτό. Είπαμε σε ποιες περιοχές θα ε, εφαρμόσουμε αυτή τη νέα συνοχή. Και εγώ είπα ότι πρέπει να την εφαρμόσουμε σε όλες για να μην υπάρξουν Νέε διαιρέσει. γιατί έτσι η Ευρώπη θα είναι πιο κοντά σε όλους τους ε, πολίτες της. Ξέρετε ότι υπάρχει ε, ένα ισχυρό αντιευρωπαϊκό ρεύμα τώρα εν ώψη και των ευρωεκλογών. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτύχει αποτελέσματα. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι δεδομένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες είχαμε την εκδήλωση με τον πρόεδρο Γιούγκερ. Είδατε πόσοι νέοι που εποφελούνται από το πρόγραμμα Έρασμος και κινούνται και για να εργαστούν από χώρα σε χώρα, αυτοί θεωρούν ότι όλα αυτά είναι δεδομένα. Δεν θυμούνται την προηγούμενη περίοδο. Αλλά κοιτάξτε, 30 χρόνια δεν είναι και τόσο πολύ στο παρελθόν. Όλοι, δηλαδή, ε, πολλοί είμαστε αρκετά μεγάλη ηλικία για να θυμούμαστε την περίοδο του κομμουνισμού που δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία επιλογή. Πού να πάμε, τι να σπουδάσουμε, πού να δουλέψουμε. Αλλά είμαστε επίσης ε, παρκώς νέοι για να αισθανόμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον των μελλοντικών γενεών. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να είναι ευφιέστερη, να έχει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, χαμηλό άνθρακα, για να διατηρήσουμε τον πλανήτη για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Τα επόμενα βήματα είναι πολύ σαφή. Έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, αλλά και εφικτό. Σας ευχαριστώ όλους που δεσμευθήκατε για αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα και ελπίζω να ξεκινήσουμε σύντομα τις διαπραγματεύσεις. Για το επόμενο πολιτές πλαίσιο υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε γύρω στους 50 τριμερείς διαλόγους. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί παίρνουν πολύ χρόνο. Εδώ είμαστε φίλοι όλοι. Γι' αυτό σας τα λέω στα ράτα και χήμα. Είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, αλλά το χαιρετίζω αυτό. Αλλά ίσως χρειάζεται να είμαστε και πιο φιλόδοξοι. Και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις και προσβλέπω και στην περαιτέρω συζήτηση και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Θα συνεχίσουμε τώρα τη συζήτηση μεταξύ των συντονιστών και των δύο επιτροπών και μετά από αυτό θα δώσω το λόγο στα μέλη και των δύο επιτροπών. Θα αρχίσουμε με τον συντονιστή από την ομάδα του ΑΕΛΚ. Είστε έτοιμος να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Ρημών θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω χωρίς προετοιμασία γιατί λείπει ο κύριος Φανίστερ. Καταρχάς ευχαριστώ τους ομιλητές γιατί είναι λυσαλέοι υποστηρικτές της ε, πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φέτος το 18 που είμαστε και στο πλαίσιο των ευρωκλογών του Μαΐου 19. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουμε. Πολύ σημαντικό. Δεν ε, εκφράζω μόνο μία ομάδα αλλά και έναν εισηγητή λέγοντας ότι τους τελευταίους μήνες κάναμε αυτό που μας είχε ζητηθεί, αυτό που ήταν σημαντικό, δηλαδή οι εκθέσεις αυτές να υποβληθούν τάξιστα στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στις Επιτροπές, ούτω ώστε να ξεκινήσει τάχιστα στο μέτρο του δυνατού ο τριμερής διάλογος. Δεν ήταν και τόσο απλό. Οι συγητές ε, ξέρουν πολύ καλά γιατί ξέρουν και πώς χρειάστηκε να εργαστούν κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Και μη πλέον δυσχέρεια είναι ότι αν μια νομοθετική έκθεση συνδέεται και με το πολιτές πλαίσιο, χρειάζεται πολύ χρόνος για να συζητήσει κανείς με όλους. Και στις ε, διάφορες περιφέρειες θα έπρεπε να έχουμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με όλους και λόγω τη στενότητα χρόνου δεν ήταν δυνατόν, αλλά κάναμε μια προσπάθεια να συναντηθούμε με του σημαντικότερου εμπλεκομένου. Και νομίζω ότι γι' αυτό προέκυψαν καλέ προτάσει που τώρα συζητούνται στι επιτροπέ και σύντομα θα πρέπει να γίνουν ε, συμβαστικέ προτάσει για όλα αυτά τα θέματα οι οποίε ε, θα αλλάξουν κάπω ε, τις προτάσεις της Κομισιόν αλλά θεωρώ ότι θα σεβαστούν τη φιλοσοφία και την βασική κατεύθυνση της ε, πρόταση της Κομισιόν και πιστεύω ότι θα τα επιτύχουμε και εγκαίρως στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει, ότι μέχρι τέλος του χρόνου δηλαδή, ίσως θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Αλλά πρέπει να θέσουμε ένα θεμελιώδες ερώτημα. Σήμερα, στις 9 Δεκάτου 18. Το θέμα είναι γιατί χρειαζόμαστε σήμερα την περιφερειακή πολιτική. Και η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο. Περισσότερο από ποτέ. Γιατί η συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο λέει πρέπει να κάνουμε περικοπές. Και ότι πρέπει το πλαίσιο αυτό πρέπει να το δέχονται και τα κράτη-μέλη. Και πάντα, όταν συζητιέται το δημοσιονομικό πλαίσιο, πάντα το πρώτο θύμα των περικοπών είναι η περιφερειακή πολιτική. Καταφέραμε την προηγούμενη φορά να διατηρήσουμε πάνω κάτω το επίπεδο, αλλά τώρα που έχουμε και το Brexit, θα πρέπει να γίνουν κάποιες περικοπές. Και το θεμελιώδες είναι ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε με την περιφερειακή πολιτική ή τι δεν θα κάνουμε εάν υπάρξουν υπερβολικέ περικοπέ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια πολύ ουσιώδη συζήτηση από αυτού λόγω τη συγκυρία. Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να διατηρηθεί ω έχει. Και αυτό για τρει απλού λόγου. Πρώτον, στην Ευρώπη η λέξη αλληλεγγύη δεν έχει πλέον την αξία ε, που τις είχαν αποδώσει οι ιδρυτικοί πατέρες και η επόμενη γενιά, ότι οι ισχυρότεροι βοηθούν τους ασθενέστερους. Αυτή είναι η βασική αντίληψη της περιφερειακής πολιτικής. Αυτή πρέπει να υπερασπιστούμε, να διατηρήσουμε και να διαμετρηθούμε αν κάποιος λέει δεν χρειάζεται πλέον. Εάν δεν υπερασπιστούμε αυτήν την αρχή, τότε η Ευρώπη χάνει την ψυχή της. Και δεν θα πρέπει να τη Γιατί εδώ είμαστε ε, περιφερειακή πολιτική και Επιτροπή Περιφερειών δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοια πράγματα. Δεύτερο λόγο. Έχει αλλάξει ο κόσμο. Και οι διαθροτικέ πολιτικέ πρέπει και αυτέ να αλλάξουν στόχου. Δεν είναι θέμα τώρα να χτίσουμε απλώ ένα αυτοκινητόδρομο. Πρέπει στο μέλλον να επενδύσουμε για αυτήν την ευφιέστερη Ευρώπη. Και όταν λέω ευφιές, smart, αυτό σημαίνει ότι μια Ευρώπη η οποία ε, είναι στην πρώτη γραμμή και θα πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή για τι καταπολέμηση κλιματική αλλαγή. Και την προηγούμενη φορά νομίζω το είχαμε καθορίσει πολύ σωστά. Πώ πρέπει να δαπανηθούν οι πόροι για την περιφερειακή πολιτική συγκεκριμένα. Και πρέπει να παίξει πρωτοπόρο ρόλο αυτή η πολιτική και πρέπει να διατηρήσει. Δημιουργούμε το μέλλον στα πλαίσια τη περιφερειακή πολιτική. Όχι απλώ επιδεικνύουμε αλληλεγγύη, αλλά διαμορφώνουμε και το μέλλον. Ποιο άλλο μπορεί να το πει αυτό. Εμεί μπορούμε να το κάνουμε. Και πρέπει να, και να το λέμε. Αλλά το λέμε ψιθυριστά. Πρέπει να το φωνάζουμε. Αυτά είναι προγράμματα που θα διατηρήσουν ε, τον κόσμο για το μέλλον των παιδιών μα. Πρέπει να το πούμε. Και κάτι που με ανησυχεί τώρα. Αλλά είναι σημαντικό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι στα κράτη-μέλη αναπτύσσεται κάπως η τάση όλο και περισσότερο ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ε, τον πρώτο ρόλο. Αυτό το America First όλο και περισσότερο ακούγεται και στα δικά μας κράτη-μέλη. Ότι πρέπει ίσως περισσότερο να ε, κλειστούμε στον εαυτό μας και να χάσουμε από την ε, οπτική μας τους γείτονές μας. Το βλέπω αυτό και στην Ιντερέγκο που είμαι εισηγητή. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα ευγενέστερο να έχουμε τρει-τέσσερι εταίρου από τρία-τέσσερα κράτη-μέλη να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να ε, καταλήξουν σε μια κοινή λύση για ένα κοινό πρόγραμμα. Έτσι έχει μέχρι τώρα λειτουργήσει η Ευρώπη ως νέος. Έτσι θα ήθελα να συνεχιστεί μέχρι να μπω σε οίκο ευγυρία. Θα ήθελα τρία-τέσσερα κράτη-μέλη να συνεργαστούν. Αυτό εκφράζει μια θεμελιώδη αξία της Ευρώπης, ότι θέλει να καταργήσει τα σύνορα. Εγώ περνάω από πολλά σύνορα και δεν το καταλαβαίνω καν πλέον. Και αυτό είναι με μια ε, βελτίωση που πολλές γενιές ούτε να την ορεινευτούν δεν μπορούσαν. Και την τάση την αντίστροφη να δημιουργούνται και να υψώνται και πάλι σύνορα πρέπει να την καταπολεμήσουμε μέσω της περιφερειακής πολιτικής. Μέσω αυτής της κοινή διαχείρισης. Shared management. Οι περιφέρειες που συμμετέχουν σε μια εταιρική σχέση να μπορούν να συνεργάζονται. Αυτό πρέπει να το περασπιστούμε. Είναι σωστή πολιτική. Είναι λογική πολιτική. Μόνο έτσι μπορεί και αύριο η Ευρώπη να συνεχίσει να λειτουργεί. Όλα τα άλλα είναι λάθος. Εάν δεν τα καταφέρουμε για αυτούς τους τρεις τομείς που τόσο έντονα τόνισα να υπάρξει η επαρκή χρηματοδότηση μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Αν βασιστούμε σε ε, έντονες περικοπές δεν θα κάνουμε τίποτα. Αλλά όσα λέμε χρειάζονται και επαρκή χρηματοδότηση. Βέβαια, εντάξει, ε, πρέπει να κάνουμε έκκληση, όχι εδώ, γιατί όλοι εδώ είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε έκκληση προ τα κράτη-μέλη. Να του πούμε, αν θέλετε αυτήν την περιφερειακή πολιτική που είναι τόσο σημαντική για του τρει προαναφερθέντε λόγου, τότε πρέπει να υπάρξει και επαρκή χρηματοδότηση. Σε τελευταία ανάλυση, εσά το ωφελεί. Πρέπει να είναι μια έκκληση προ όλου που εργάζονται σε αυτή την πολιτική να ασκήσουν πίεση στα κράτη-μέλη, ώστε τα κράτη-μέλη να προβλέψουν επαρκεί χρηματοδοτήσει. Προκύπτει και από τη δική μου έκθεση για το Interreg. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να κάνουμε και την καλύτερη ε, διαφήμιση για την Ευρώπη. Εάν θα έπρεπε να αναθέσουμε σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων να κάνει ε, διαφημιστικές ε, εκστρατείες για την Ευρώπη, αυτά θα τους δίναμε θα του λέγαμε ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσετε την Ευρώπη είναι η περιφερειακή πολιτική. Παρουσιάστε την καλύτερα. Πείτε ότι η Ευρώπη συγχρηματοδοτεί υποδομές, ε, ε, πόλου, ευφυείς πόλεις, ε, νοσοκομεία. Θα καταλάβουν οι πολίτες πόσο σωστή είναι η Ευρώπη. Βεβαίως και μέσω του κανονισμού Omnibus προβλέπουμε χρηματοδοτήσεις και ακριβώς για τέτοιες διαφημιστικές εκστρατείες για την Ευρώπη. Οι εμπλεκόμενοι στην ε, περιφερική πολιτική θα πρέπει και αυτοί να πιστούν ότι και αυτοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν. Μία επιχείρηση, μία ΜΚΟ, οποιοδήποτε έχει συμμετάσχει στα προγράμματά μας να έχει την εντύπωση ότι είναι καλύτερα να πάει σε τράπεζα για να χρηματοδοτηθεί και όχι να ζητήσει χρηματοδότηση γιατί είναι περίπλοκη η διαδικασία. Αυτή ήταν μέχρι τώρα η τάση. Πρέπει να την αντιστρέψουμε τόσο ώστε όλοι να θέλουν να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους μέσω κοινή διαχείρισης. Αν το επιτύχουμε αυτό, δεν θα προωθήσουμε μόνο την ε, περιφερειακή πολιτική, αλλά και συνολικά την Ευρώπη. Θα εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη. Άρα θα εξυπηρετήσουμε και όλους μας. Θα επιτύχουμε κάτι και σημαντικό και καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα από την Επιτροπή των Περιφερειών, η Κατιούσα Μαρίνη είναι συνεισηγήτρια για τον κανονισμό περί διατάξεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε της Επιτροπής ε, Ρέτζιε και αγαπητή κυρία Επίτροπε. Πιστεύω ότι αυτή η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική για τις εργασίες μας και από την πλευρά της Επιτροπής των Περιφερειών και ιδιαίτερα από την οπτική των περιφερειών και των πόλεων γιατί εμείς είμαστε πρόσωποι και διοικητές αυτών των ε, περιοχών. Το θέμα το, του μέλλοντος της πολιτικής συνοχής ε, δεν είναι μόνο, όπως πολύ σωστά υπογράμμισε η Επίτροπος, ε, η κυριότερη πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συγκεντρώνονται πόροι και όπου ερμηνεύεται όπως υπόθηκε ήδη η ιδέα της αλληλεγγύης και της ε, διαδικασίας ε, ολοκλήρωσης και ξεπεράσματος των ανισοτήτων αλλά η πολιτική αυτή για τις περιφέρειες και τις πόλεις είναι ε, το κύριο, η κύρια πολιτική στρατηγικών επενδύσεων και θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι. Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και στις πόλεις των κρατών μελών, που ε, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης των, ε, της δημοσιονομικής και του εθνικού χρέους, ε, πολύ συχνά η πολιτική συνοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η μόνη πολιτική στρατηγικών και διαρθρωτικών επενδύσεων που διέθεταν αυτές οι κοινότητες. Και έτσι οι διαχειριστές των πόλεων αυτών και των περιφερειών κατάλαβαν σε βάθος όχι μόνο τη σημασία αλλά και τη δύναμη αυτής της πολιτικής. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί θεωρούμε ότι ε, έχοντας μπροστά μας την πρόταση της Κομισιόν αλλά και διαπραγματεύσεις σημαντικές ότι θα πρέπει να χτιστεί μια ε, πολύ σημαντική συμμαχία ανάμεσα στην ε, ε, Επιτροπή των Περιφερειών και την Επιτροπή Ρέτζη γιατί η Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπεί πιο άμεσα ε, τις ε, περιφέρειες και τις πόλεις και το Κοινοβούλιο από την άλλη πλευρά είναι η άμεση έκφραση της φωνής των πολιτών αλλά και η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει την, τους τοπικούς φορείς, τις τοπικές κοινωνίες. Όλα αυτά για να αποφύγουμε ένα πράγμα. Να μην γίνεται αντιληπτή η πολιτική ε, συνοχής ε, ε, αντιληπτή μόνο σαν ένα σωσίβιο για τις περιφέρειες και τις πόλεις που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες μέσα στην Ευρώπη, αντίθετα να γίνεται αντιληπτή σαν μια διαρθρωτική πολιτική που να αφορά με στρατηγικό τρόπο όλες τις περιφέρειες, όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Και γι' αυτό συμφωνούμε απολύτω με το σημείο αυτό τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχή σε μια πολιτική για όλου. Για να προωθηθούν οι επενδύσει, η καινοτομία, η ανάπτυξη που αφορά αυτό όλε τι περιφέρειε, όλε τι περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο τι λιγότερο ανεπτυγμένε. Θα θέλαμε επίση να επαναλάβουμε το γεγονό ότι Κάτι τέτοιο θα πρέπει να διατηρήσει ένα χαρακτήρα ε, τοπικής και τοπικού και περιφερειακού προγραμματισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που υπάρχει στο σημερινό πλαίσιο ε, που ε, συνδυάζεται με την αρχή της επικουρικότητας, με την συμμετοχή των θεσμικών εταίρων αλλά και κοινωνικών και οικονομικών εταίρων στον προσδιορισμό αλλά και στην υλοποίηση των ε, ε, πολιτικών που βασίζονται στην πολιτική συνομνοχή και στο σχετικό προγραμματισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην έκθεση, στη γνωμοδότηση, συγγνώμη, ε, που ετοιμάζουμε, διότι τον Οκτώβριο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κοτέρ. Εγώ και ο Συνάδελφο Βάιντερ τονίσαμε πάρα πολύ την ανάγκη να αποφύγουμε ορισμένα κράτη-μέλη να οθήσουν προς μια αξιοποίηση ουσιαστικά ε, συγκεντρωτική σε εθνικό επίπεδο των πολιτικών αυτών ε, σε υποκατάσταση των ε, εθνικών δαπανών προς τις περιφέρειες. Εμείς στην ουσία θέλουμε η πολιτική αυτή να είναι ένα εργαλείο στη διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις και τις επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας. Και γι' αυτό συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά ε, τον ορισμό των περιφερειών ε, σε φάση μετάβασης και από αυτό θα θέλαμε να ε, τονίσουμε δύο σημεία και, σε με αυτό θα τελειώσω. Ε, λέω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε περαιτέρω σημεία σύγκλησης. Δεν εστιάζω μόνο ε, στα σημεία που μας βρίσκουν σύμφωνους, ίσως ε, αντίθετα θα ήταν σημαντικό να συζητήσουμε αυτό ε, που ανέφερα πριν, δηλαδή και στην Επιτροπή Ρέτζι να ε, υιοθετηθεί η άποψη να δοθεί εστίαση στο προγραμματισμό σε τοπικό επίπεδο για μας είναι σημαντικό να ε, προωθηθεί η έννοια τη απλούστευσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να φτάνει στου πολίτε, στις επιχειρήσει, ακόμα και στι πιο μικρέ τοπικέ και περιφερειακές διοικησει. και άρα οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε δεν πρέπει να είναι φραγμός, δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για τη χρήση αυτού του εργαλείου. Όσο πιο εύκολη είναι η πρόσβαση στην, στην πολιτική συνοχή, τόσο πιο πολύ η Ευρώπη θα αποδειχθεί ότι στέκεται κοντά στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και έτσι θα έχουμε ε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες και αυτό φαίνεται και στην ε, γνωμοδότησή μας σχετικά με την επανεισαγωγή του κανόνα νησιν 2. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο για τις τοπικές αρχές να παραμείνει ενισχύει ο σημερινός κανόνας νησιν συντρία για να αποφύγουμε και προβλήματα προγραμματισμού γιατί βρισκόμαστε σε ένα και κεκαιώνα επικάλυψης ανάμεσα στην παλιά, στον παλιό ε, προγραμματισμό που μπορεί να ε, πειράσει όλες τις ε, περιοχές όπου εστιάζονται περισσότερο οι στρατηγικές επενδύσεις και θεωρούμε ε, το είπατε αυτό στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι σκέφτεστε από αυτού. Για μας όμως είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να εξαρτάται από μακροοικονομικούς όρους που δεν ε, ε, είναι στην αρμοδιότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά θα μπορούσαν να ήταν σημεία σύγκληση ε, μεταξύ μα. Είναι σημεία τα οποία τονίζουμε στην γνωμοδότησή μα και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική και στρατηγική δουλειά για να διασφαλίσουμε όχι μόνο μια πολιτική αλλά και μια ιδέα της Ευρώπης απέναντι στις ε, περιφέρειες και ε, η ισχυρή πολιτική συνοχής είναι ένα από τα πιο χειροπιαστά και αναγνωρίσιμα πράγματα του τι είναι η Ευρώπη ε, όσον αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση, τις πολιτικές εργασίες, τις στρατηγικές επενδύσεις, το περιβάλλον, τις ε, ε, επενδύσεις στο αστικό περιβάλλον και σε όλα αυτά η Ευρώπη βοήθησε όχι μόνο οικονομικά, αλλά με μια κουλτούρα ε, πολιτική, μια ε, κουλτούρα προγραμματισμού ε, που σε πολύ υψηλό επίπεδο εμπλέκονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εν ώψη του 2019 εδώ παίζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης της Ευρώπης σε σχέση με τους πολίτες. Δεν μπορούμε κατά κανένα τρόπο να υποθέσουμε και αυτό θα το πούμε και στις διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ότι δεν θέλουμε η η λογική της περικοπής των προπολογισμών να μας φέρει σε μια επανεθνικοποίηση των πολιτικών αυτών και ε, στο σημείο αυτό είμαστε εντελώ αντίθετοι και στη γνωμοδότηση το τονίζουμε πάρα πολύ το σημείο αυτό θα ήμασταν εξάλλου ε, ε πρόθυμοι να ε, υπερασπιστούμε τη θέση αυτή και σε εθνικό επίπεδο, ότι δηλαδή όχι μόνο θα πρέπει ε, τα κονδύλια να, είναι, ε, να μην περικοπούν, αλλά να εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κρέλ, που είναι η συντονίστρια των σοσιαλιστών. Ε, στην Επιτροπή Ρέτζη, αλλά και η εισηγήτρια για τον ε, CPR. CPR. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Αϊμού για την πολιτική συνοχή. Συμφωνούμε απόλυτα. Συνυπογράφω. Οπότε και δεν θα επαναλάβω. Αλλά να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη όπως και η Επιτροπή Περιφερειών έναντι των ε, συμπολιτών μας. Γιατί είμαστε η άρθρωση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών γενικά οτιδήποτε και αν ε, σημαίνει αυτό και από την άλλη μεριά των ε, πολιτών. Είμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές και είμαστε βεβαίως τμήμα και εμείς των ευρωπαϊκών θεσμών. Και ακριβώς για την πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η πολιτική συνοχή είναι το μόνο επενδυτικό μέσο το οποίο συναποφασίζεται με τις περιφέρειες και τις πόλεις και τους δήμους όπου ακριβώς υλοποιείται αυτή η προσέγγιση ότι αυτά που θα ε, εφαρμοστούν επιτόπου αποφασίζονται και επιτόπου με τα χρήματα των Ευρωπαίων ακριβώς, ακριβώς φορολογουμένων. Γι' αυτό τη χρειαζόμαστε και στο μέλλον. Στα κράτη-μέλη αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός. Πολλές κυβερνήσεις ε, υφίστανται ισχυρούς πειρασμούς επανεθνικοποίησης των πολιτικών. Ξέρουμε, όλοι που είμαστε εδώ, ότι αυτό δεν θα αποτελέσει επιτυχία για την Ένωση. Πρέπει όντως και πάλι να δημιουργήσουμε πνεύμα εμπιστοσύνης στους πολίτες ότι οι καλύτερες λύσεις προκύπτουν μέσω της Ένωσης. Και γι' αυτό τον λόγο η πολιτική συνοχής δεν πρέπει μόνο να επενδύσει σε συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά να επενδύσει και για να υπάρξει ή να επανέλθει το κλίμα εμπιστοσύνης προς την Ένωση. Τι πρέπει να κάνει η Ένωση ε, σε έναν κόσμο ο οποίος γίνεται όλο και πιο περίπλοκος που αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά νομίζω μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Βεβαίω ξέρω ότι πρέπει να απευθυνθώ σε αυτού που δεν είναι εδώ παρόντε, αλλά ίσω να μα ακούσουν παρόλα αυτά. Θέλω λοιπόν να υπάρξει έκκληση όσο πιο σύντομα και με βάση και τα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο δυνατόν πιο κοντά δηλαδή, να καθοριστεί το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ω Επιτροπή έχουμε δεσμευθεί όσο ταχύτερα γίνεται να υπάρξει εντολή για τους κανονισμούς ε, της η πρόεδρος το είπε στην αρχή. Το Δεκέμβριο θέλουμε να αποφασίσουμε για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις του τριμερούς διαλόγου. Θα το επιτύχουμε και για τον συνολικό κανονισμό. Νομίζω ότι με τον συνεισηγητή μου Αντρέι Νόβακοφ θα τα καταφέρουμε. Να ξεκινήσουν δηλαδή οι διαπραγματεύσεις. Στόχος μας είναι, τουλάχιστον όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη διαχείριση, να διεξαχθούν οι διάλογοι και να ολοκληρωθούν, ούτω ώστε να γνωρίζουν οι περιφέρειες τι θα προκύψει. Γιατί είναι τρομερά σημαντικό. Αλλά από πάνω μας πάντα επικρέμαται η δαμόκλειος σπάθη του αποτελέσματος ε, των διαπραγματεύσεων του ΠΔΛΤΑΠ. Δεν υπάρχει συμφωνία για τις προτάσεις του Έτινγκα και δεν υπάρχει και συμφωνία για το τι θέλει το Κοινοβούλιο. Δηλαδή τι μπορεί να συμβεί αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει επί περικοπών επί της προτάσεως της Κομισιόν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ξαναδούμε συνολικά την πολιτική συνοχή. Εγώ δεν το θέλω. Και γι' αυτό πρέπει να στείλουμε το μήνυμα από αυτή την κοινή μας συνεδρίαση προς το Συμβούλιο ούτως ώστε να υπάρξει μια συμφωνία κάπου μεταξύ των προτάσεων ε, Επιτροπής και Κοινοβουλίου για να έχει έννοια η περαιτέρω εργασία μας. Τι προτείνουμε στα πλαίσια αυτού του συνολικού κανονισμού. Η Επιτροπή, και την ευχαριστώ, κάνει πρόταση να συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες στην συνοχή. Γι' αυτό είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Είναι θεμελιώδης απόφαση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αλλά η πολιτική συνοχής στο μέλλον θα πρέπει να εργάζεται με πολύ στενή συνεργασία με τις περιφέρειες, με την τοπική αυτοδιοίκηση και κατά τη φάση προετοιμασίας. Αυτό θα το τονίσουμε ακόμη περισσότερο. Επίσης, είναι σημαντικό η ανάπτυξη της υπαίθρου να ληφθεί υπόψη περισσότερο, να συμπεριληφθεί. Και όχι η ανάπτυξη της υπαίθρου να προωθείται μόνο μέσω της ενίσχυσης των γεωργών. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να το συνδέσουμε μέσω αυτού του γενικού κανονισμού. Και γι' αυτό η Επιτροπή μας προτείνει το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου να υπαχθεί και πάλι σε αυτόν τον γενικό κανονισμό. Όπως είπε και ο συνάδελφος Αριμό, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα το πρόγραμμα Interreg να λάβει περισσότερη, ουσιοδός περισσότερη χρηματοδότηση. Και γι' αυτό προτείναμε στην Ρέγγι να αυξηθούν κατά 3% οι πόροι του Interreg. Και θα πρέπει να δούμε ότι αυτό θα αυξήσει την ορατότητα και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ούτω ώστε να υπάρχει περισσότερη συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Επίσης, από την άλλη πλευρά, οι πόροι που θα έχουμε στη διάθεσή μας να συνδυάζονται πιο αποτελεσματικά και απλούστερα με άλλα προγράμματα της Ένωσης. Και αυτό το θεωρούμε σημαντικό. Και θέλω να πω σαφές, σαφώς ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς ένα μέσο για να κάνουμε κάπου και κάπως επενδύσεις. Η πολιτική συνοχής είναι ένα μέσο που θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την έρευνα και καινοτομία, με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή ε, είναι, ανοιχτό, είναι ανοιχτή η πολιτική συνοχής προς το μέλλον περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέσο της Ένωσης. Και γι' αυτό πρέπει να συνδεθεί σωστά και με το μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας Horizon Ευρώπη και με το πρόγραμμα InvestEU που είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα συζητήσουμε αν θα συμφωνήσουμε σε μεταφορές πιστώσεων. Οι εισηγητές ε, το απορρίπτουν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από αυτού. Το επόμενο διάστημα θα επιτύχουμε σίγουρα, θεωρώ, συμβασμούς. Εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου προς την Κομισιόν για το πόσο μα στήριξε για να επιβληθεί στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus απλούστευση των διαδικασιών ούτω ώστε να υπάρξει κατόπιν ε, απλούστευση και των περαιτέρω κανονισμών. Το υποστηρίζουμε αυτό. Δεν έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία σε αυτή τη ε, διαμόρφωση να συζητήσουμε με την Επιτροπή Περιφερειών. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παράκληση προς τις περιφέρειες δεν έχει έννοια η απλούστευση να γίνεται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απλούστευση και η συνεργασία για να εφαρμοστούν οι προτάσεις που υποβάλλει η Κομισιόν πρέπει να υπάρχουν λοιπόν αυτά και σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο περιφερειών. Και τα ξέρω πολύ καλά. Πολύ συχνά επισκέπτομαι διάφορες περιφέρειες και όχι μόνο πραγματικά πιστέψτε με όχι μόνο γερμανικές περιφέρειες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ιστερήσεις στα κράτη-μέλη ούτως ώστε να υπάρξει απλούστευση κάθε κράτος μέλος δηλαδή στο εσωτερικό το δικό του και δεν μας βοηθάει αν μετά από πέντε χρόνια έρθουμε πάλι και πούμε θέλουμε όλα να είναι απλά αλλά αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες φταίνε που δεν λειτουργεί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι θα το πληρώσουμε. Γιατί έτσι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ευρωσκεπτικισμός. Πρέπει όλοι τώρα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να υπάρξει απλούστευση σε όλα τα επίπεδα. Σας παρακαλώ να το ε, μεταφέρετε αυτό παντού και στις περιφέρειές σας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μόνο στη δική μας λειτουργία πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη για να προχωρήσουμε όλοι από κοινού. Και αυτό θα το αναφέρουν πολύ περισσότερο οι εισηγητές του Γενικού Κανονισμού. Θέλουμε καλύτερη πολιτική ενημέρωση. Εάν δαπανούμε από κοινού πόρους να εφαρμόζονται για προγράμματα που να έχουν έννοια. Και πολλοί πολίτε δεν έχουν ιδέα για το πόσα επενδύει η Ευρώπη στην περιφέρειά τους. Ας ε, θυμηθώ τις διαπραγματεύσεις για τον προηγούμενο γενικό κανονισμό. Ένα από τα πιο δυσχερή θέματα κατά τον τριμερή διάλογο ήταν του πώς θα βάλουμε μια ταμπέλα που να λέει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εν τω μεταξύ έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Για παράδειγμα, εάν ε, στο, σε ένα γραφείο του Οργανισμού Ευρέσεως Εργασίας, για παράδειγμα, βάλουμε μια πινακίδα που να λέει ότι εδώ μπορείτε να συμμετάσχετε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι πολλοί έχουν αντιρρήσει βεβαίω ότι όχι, εδώ είμαστε ένα οργανισμό, δεν μπορούμε να βάζουμε πινακίδε που να λένε ότι να είναι. Πρέπει να υπάρχει όμω αυτό. Ούτω ώστε να εγκαταστεί σαφέ ότι η Ευρώπη συμμετέχει στην εξέβρεση λύσεων στι περιφέρειε για του πολίτε. Και πρέπει να λέγεται αυτό, πρέπει να αναφέρεται. Πιστεύω του επόμενου μήνε, όχι κατά την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και ευρύτερα είναι αναγκαίο να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είμαστε πολύ πιο παρόντες και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε σε θέση να βρίσκουμε και να εφαρμόζουμε λύσεις. Να μην ε, μας παρουσιάζουν ως τμήμα του προβλήματος. Η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα. Η Ευρώπη είναι η λύση για το μέλλον και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ε, εργαστούμε πολύ περισσότερο για να επιτύχουμε από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μιχάλης Σνάιντερ, ο συν, ε, ε, για τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, χρειάζεται και να τονίσω πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κανονισμός. Νομίζω ότι η ανταλλαγή απόψεών μας πάντα έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα που έχουν θετικέ θετικές επιπτώσεις για όλη την Ένωση. Δεν υπερβάλλω που το λέω. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που όλοι κερδίζουμε. Εσείς ε, συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα αιτήματά σας. Και εσείς μαθαίνετε βεβαίω επίσης από εμά πώς εφαρμόζεται η πολιτική συνοχή. Εμείς την εφαρμόζουμε και μπορούμε να σας δώσουμε ουσιώδη στοιχεία για το τι πάει καλά και τι όχι. Δηλαδή, εποφελούμεθα και οι δύο από τέτοιε συναντήσεις. Γι' αυτό ευχαριστώ και πάλι. Δεν θα πω κι εγώ πόσο πιστεύω στην πολιτική συνοχή. Ε, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ αυτά. Γιατί ήδη έχουν ε, υποθεί πολλά. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Συμπληρώνοντας ε, τα συγκεκριμένα που και εσείς βεβαίως είπατε. Να σας αναφέρω ένα παράδοξο. Την περασμένη εβδομάδα λάβαμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το ποσοστό σφαλμάτων για την εφαρμογή των διαθροτικών ταμείων. Μειώνονται όλο και περισσότερο. Είναι κάτω από 3%. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες ε, είδαμε στον τύπο ότι τα ποσοστά εκταμίευσης των διαθροτικών ταμείων δεν είναι τα βέλτιστα. Τι γίνεται, πού οφείλεται αυτή η διαφορά και τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί η απορρόφηση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την πύρα της προηγουμένης ε, περίοδου για την επόμενη περίοδο. Έχουν ήδη γίνουν κάποιες προτάσεις. Το σημαντικότερο είναι η διοικητική απλούστευση. Πάντα στις γνωμοδοτήσεις μας ε, το τονίζαμε τα τελευταία χρόνια το θέμα αυτό. Και έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Κρέτσου. Δεν πρέπει να κατηγορούμε μόνο τις Βρυξέλλες. Πρέπει και εμείς αυτοκριτικά να δούμε πώς λειτουργεί η κάθε περιφέρεια. Εγώ συμμετέχω στην διοίκηση μιας περιφέρειας. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας. Ούτω ώστε να απλουστευτεί η κατάσταση για την επόμενη περίοδο. Και αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν επαρκεί κάτι μας. Η γνωμοδότηση που θα αποφασίσουμε στην Ολομέλειά μου στο Δεκέμβρη, Μαρίνη και δική μου, θα περιέχει πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Από την πείρα μα. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει περαιτέρω διοικητική απλούστευση. Πώς τώρα μπορούμε να βελτίσουμε την απορρόφηση για να το βοηθήσουμε αυτό πρέπει να υπάρχει δικαιότερη κατανομή των πόρων. Γιατί έχουμε τρεις ε, κατηγορίες περιφερειών. με βάση τις οποίες κατηγορίες ε, καθορίζονται και οι όγκοι. Αλλά προβλέπονται ε, ε, σοβαρές μειώσεις της χρηματοδότησης και αυτό μας ανισχύει ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες σε μετάβαση. Η Κομισιόν προτείνει μείωση από το 80% στο 55%. Εσείς από ό,τι ακούω θέλετε να προτείνετε 60%. Στην χρηματοδότησή μας προτείνουμε 70%. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ε, καθημερινής μου πείρας. Εγώ ε, είμαι από μια μεταβατική ε, μια περιφέρεια σε μεταβατική φάση. Αν μειώσουμε κατά 20-25% τη συγχρηματοδότηση, θα έχουμε μεγάλες δυσχέρειες για να απορροφήσουμε διαφορετικούς πόρους. Έχουμε όλοι ε, πολύ ισχυρή δημοσιονομική πειθαρχία στις περιφερειές μας που πρέπει και θέλουμε να τηρήσουμε. Γιατί χρειάζεται τέτοια πειθαρχία για να αποφεύγεται η ε, σπατάλη. Δεν είναι τόσο μεγάλο, η μεγάλη Το μεγαλύτερο τμήμα των προπολογισμών μας είναι υποχρεωτικέ δαπάνε. Δεν έχουμε πολύ περιθώριο χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων. Αν μας μειώσετε τη χρηματοδότηση θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η απορρόφηση των διδακτικών πόρων. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεύτερο σημείο. Κατανομή των πόρων, όπου δεν συμφωνούμε ακόμη. Πολύ καλή ιδέα, κυρία Κρέτσου, και το χαιρετίζω αυτό που είπατε. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο ασφαλείας, είπατε, ένα δίκτυο ασφαλείας. Είπατε ότι κανείς δεν θα πρέπει να χάσει πάνω από 24%. Άρα είπατε ε, ότι το δίκτυο ασφαλείας πρέπει να είναι στο 76%. Αλλά αυτό που καθορίζει το δίκτυο ασφαλείας είναι του εθνικό επίπεδο. Και σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν περιφέρειες που υπάρχουν ε, περιοχές με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξη. Εγώ είμαι την Ανατολική Γερμανία. Εάν το δίκτυο ασφαλείας είναι 76% τότε οι πιο ευημερούσε περιοχές στην ε, δυτική, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας θα χάσουν ε, λιγότερα από ό,τι θα χάσουμε εμείς στι πιο αδύναμε περιοχέ. Γι' αυτό καλό το Κοινοβούλιο να σκεφτεί την πρότασή μα και πάλι. 76% ναι, αλλά ε, το κριτήριο πρέπει να είναι το περιφερειακό επίπεδο, η σημερινή χρηματοδότηση της κάθε περιφέρειας. Στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους είναι το ουσιώδες πώς θα γίνει η κατανομή των πόρων. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό ε, αίτημα. Και να υπογραμμίσω αυτό που είπε και συνάδελφος Μαρίνη, το νήσι 2 ή νήσι 3. Ιδιαίτερα στην αρχή της νέας περίοδου προγραμματισμού, η ε, μετάβαση στον ΙΣΙΝ 2 θα δημιουργήσει ουσιώδη προβλήματα. Πρέπει να ολοκληρωθεί η τωρινή περίοδος όπου ισχύει το ΙΣΙΝ αλλά θα αρχίσει και ελπίζω ε, έγκαιρα, χωρίς να το πολύ πιστεύω, η νέα περίοδος, οπότε όλα θα πέσουν μαζί. Θα έχουμε τις ίδιες δυσχέρειες στην έναρξη της νέας περίοδου που είχαμε και στην έναρξη της προηγούμενης. Και ξέρετε, η αρχή είναι το ίμιση του παντό. Άμα ξεκινήσει άσχημα, η απορρόφηση θα συνεχιστεί και άσχημα. Αυτά είναι τα τρία σημαντικότερα σημεία όπου ακόμη υπάρχουν διαφορέ αντιλήψεων, Σα παρακαλώ. Δίκτυο σε περιφερειακό επίπεδο, συγχρηματοδότηση ιδιαίτερω για περιφέρειες μεταβατική περίοδου και συν 3 για την επόμενη περίοδο. Να διατηρηθεί παρακαλώ. Θα ήταν σημαντική η συνοχή που μπορούμε να ε, κάνουμε για να ε, υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση και επαρκής απορρόφηση για την επόμενη περίοδο. Βεβαίως ε, θέλω όλοι να επιτύχουμε όσο γίνεται για να ε, συμφωνηθεί το ΠΔΠ πριν τις ευρωεκλογέ. Συμφωνούμε απόλυτα στο πλευρό σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι αυτό είναι κρίσιμο θέμα πριν από τι ευρωεκλογέ να ληφθεί αυτή η απόφαση για τον ΠΔΛΤΑΠ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και για την κοινή μα αυτή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαν Μίλτερμπορκ που είναι συντονιστής της ε, ομάδας Άλτες στην Επιτροπή Ρέτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ευχάριστη αυτή η ευκαιρία που μα δίνεται για να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους τη Επιτροπή των Περιφερειών της προτάσεις τη Κομισιόν. Χρήσιμο. Θα είμαι σύντομο ώστε να μπορέσουν και άλλοι να κάνουν ερωτήσεις. Όπως είπα, ε, στην ίδια αυτή ομίγυρη, την ίδια σύνθεση με τη σημερινή, είπα ότι δεν χρειαζόμαστε επανάσταση όσον αφορά ε, ε, τον εξυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής αλλά την εξέλιξη και χαίρομαι που υπάρχει μια, ε, ένα ενδιαφέρον για μια μετατροπή της Επιτροπής Συνοχής με στοιχεία εξυγχρονισμού και εξακολουθούμε να καλύπτουμε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης όχι τις, τις περιοχές που έχουν ανάγκη για αλληλεγγύη αλλά πρέπει να επενδύσουμε και στις περιφέρειες οι οποίες ε, ε, είναι στο, στο, έχουν το προβάδισμα γιατί εκεί υπάρχει ανάγκη, ανάγκη εξειδίκευσης. Και βεβαίως το θέμα του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι σημαντικό. Κάθε ευρώ που ε, ξοδεύεται σήμερα για να αποφύγουμε την ε, υπερθέρμανση του πλανήτη θα μας εξοικονομήσει στο, ε, χρήματα στο μέλλον. Αν δει κανείς την έκθεση του IPCC πρέπει κανείς να καταλάβει πόσο πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Έχουμε νέα στοιχεία. Ένα από αυτά που είναι προσφυλές στις καρδιές των φιλελευθέρων είναι τα νέα στοιχεία του προγράμματος Interreg, ένα στοιχείο που θα επιτρέψει καινοτόμες διαπεριφερειακές επενδύσεις, η υποστήριξη της ομάδας των οικονομικών παραγόντων για την πραγματική υλοποίηση της ευρωπαϊκής, αν όχι και πανευρωπαϊκής ξυπνής εξειδίκευσης. Αυτό θα μας επιτρέψει εμάς στην Ευρώπη να είμαστε πρώτο πόροι στον τομέα της κοινοτομία. Δεν ε, ανταγωνιζόμαστε πάντα ο ένας τον άλλον. Μην ξεχνάμε ότι ανταγωνιζόμαστε τον υπόλοιπο κόσμο, Ηνωμένε Πολιτείε, Κίνα, άλλες χώρες της Ασίας και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και ένα σημαντικό εργαλείο. Ας ε, ε, δούμε λοιπόν τις προτάσεις αυτού, του στοιχείου. Ενδεχομένως δεν έχουν όλα σχέση με το χρήμα. Ενδεχομένως ε, δύο λόγια για τον Ευρωπαϊκό Διαμεθοριακό Μηχανισμό που επισημαίνει για την κομμάτι του πακέτου ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρηματοδότηση του Ιντερεγ για την προώθηση της διαμεθοριακής συνεργασίας. Χρειαζόμαστε απλώς μια ε, νομοθετική πρόταση όπως αυτή που έχει ε, τεθεί τώρα για να ξεπεραστούν διοικητικά και νομικά εμπόδια. Ως εισηγητής χαίρομαι που μπορώ να συνεργαστώ με τον Επιτρόπο των Περιφερειών επί της πρότασης αυτής. Πραγματικά κάνουμε τα σωστά βήματα και προ τη σωστή κατεύθυνση. Δύο λόγια όσον αφορά κάποια πολύ λεπτά θέματα. Θεωρώ ότι ε, δεν πιστεύουμε στις περιφέρειες. Γιατί θα πρέπει η πολιτική συνοχή να είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, γιατί να είναι συνδεδεμένη με τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και τέλο, γιατί πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τι δαπάνε του ευρωπαϊκού ε, ε, προπολογισμού και το σεβασμό του κράτου δικαίου. Θέλω να κάνω θερμή έκκληση. Μην ξεχνάμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούν να βελτιώσουν το κράτος δικαίου, την οικονομική διακυβέρνηση των κρατών μελών και γι' αυτό θα επηρεά... και αυτό θα επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των περιοχών μας. Ε, δεν είναι μια απομονωμένη πολιτική πολιτική συνοχή. μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ενσωματωμένη στις ευρωπαϊκές πολιτικές και είναι βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω στο μέλλον να θεωρείται μια ε, πολιτική ενταγμένη, ε, ολοκληρωμένη και να προωθεί την καλή, σωστή διακυβέρνηση στα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι ο τρόπος που μπορεί να είναι αποτελεσματική για μα όλους η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή. Και μπορούμε να επωφεληθούμε από τα αποτελέσματα αυτά στις δικές μας περιφέρειες, οπότε αν ε, εμπλακούν και τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες θα έχουμε μια καλή, ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο ερχόμενο όχι διάστημα απλώ αλλά στι μελλοντικέ δεκαετίε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εσμπερμαν, ελπίζω να είπα καλά το όνομά σας. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω σήμερα το λόγο στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Είναι σημαντικό που συνεργαζόμαστε επ' αυτού του θέματος που είναι πολύ προσφυλές στις περιφέρειες όπως ε, ακούστηκε. Είμαι εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειών για το, ε, για το Ταμείο Συνοχής και για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ERDF και θα επικεντρωθώ σε αυτά. Το επόμενο διάστημα, στο επόμενο δεκαπενθήμερο, θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησής μου στην Επιτροπή ΚΟΤΕΡ. Θα μιλήσω για το σχέδιο που δεν έχει ακόμα συζητηθεί στην Επιτροπή των Φεριών. Μην το ξεχνάστε αυτό, παρακαλώ. Συντάσσω το σχέδιο σε καλή συνεργασία με μέλη της Επιτροπής ε, Ρέτζι, τον κύριο Κοτσουλίνο και τον κύριο Βαν Κάρσελ και την κυρία Μιχαήλοβα. Είναι καλό που διαπιστώνουμε ότι ε, συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα που είναι σημαντικό για τις περιφέρειες. Κυρίως προτείνονται περικοπές στους προϋπολογισμούς. Αυτό είναι λυπηρό. Είναι θέμα που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες αρκετά, δεν θα επισέλθω λοιπόν. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για, την, έχουν γίνει από την πρόταση της DG Regio. Έχουν γίνει πολλά από της πρότασης αυτής. Έχουν γίνει θετικά βήματα που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Άρα δεν θα προτείνω δραστική ε, ε, μετακίνηση από το δρόμο που προτείνει η Κομισιόν, απλώς να επισημάνω κάποια σημεία που κάποιες βελτιώσεις θα είναι πολύ ευπρόσδεκτες. Καταρχήν, με χαρά άκουσα τους ομιλητές και την Επίτροπο να αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να μείνει πίσω οποιαδήποτε περιφέρεια. Μιλάμε για όλες τις περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες της πρέπει να ξεκινά από τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η πολιτική συνοχής είναι η πολιτική που θα φέρει πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της. Τώρα, οι προτάσεις το έχουν διατυπώσει ότι η θεματική ε, επικέντρωση σε θεματικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο, η θελούσια μεταφορά πόρων προς το πρόγραμμα InvestEU και αλλού που είναι το 5% του προϋπολογισμού και τέτοιου είδους θέματα ε, μας δημιουργούν την εικόνα ότι υπάρχει μετατόπιση από το περιφερειακό στο εθνικό επίπεδο και επειδή εγώ προέρχομαι από περιφέρεια, ε, το θεωρώ ε, κρίμα. Είναι ε, μια πρόταση επί της οποίας θα προτείνουμε τροπολογίες. Στις συνομιλίες μου με τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο κατάλαβα ότι αυτή η μετατόπιση από το περιφερειακό στο εθνικό επίπεδο έγινε, δεν έγινε σκόπιμα. Οπότε ελπίζω ότι θα κριθούν οι προτάσεις μας ε, κατά, τον ίδιο τρόπο, κατά αυτόν τον τρόπο από την Κομισιόν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε βήματα προς την περιφερειοποίηση της πολιτικής συνοχής ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πράγματι πιο κοντά στους πολίτες της. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ε, το κοινωνικό σκέλος του ERDF. Ε, προτείνουμε ε, τροπολογίες για την κατάργηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων. Αυτά νίκουν ήδη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά δεν επαναλαμβάνονται στο ERDF και είναι πολύ σημαντικό να επιγραμμίζουμε τα θέματα αυτά όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλο σκέλος ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και θα έλεγα στον τίτλο των πιο κοινωνικών θεμάτων εμπίπτουν και τα δημογραφικά ζητήματα ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει ε, εγκατάλειψη τον πληθυσμό, γιατί γίνεται μετανάστευση εντός της Ένωσης. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην μετανάστευση προς την Ένωση, αλλά και η εσωτερική μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα, λύνει και προβλήματα ενδεχομένως, αλλά μπορεί το θέμα αυτό να ενισχυθεί στον κανονισμό του ERDF. Επίσης θα προτείνουμε τροπολογίες ώστε ο κανονισμός να γίνει πιο πράσινος. Φυσικά είναι ένας από τους στόχους της πολιτικής, η Ευρώπη να γίνει πιο πράσινη. Πρέπει όμως να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ε, να κινηθούμε συγκεκριμένα προς θέματα που αφορούν ε, το κλίμα, την φυσική προσαρμογή, τους, τις φυσικές καταστροφές. Είδαμε φυσικές καταστροφές ε, τα τελευταία χρόνια, πλημμύρες και σεισμούς και άλλα. Θα ήταν καλό να υπάρχουν πόροι που να κινηθούν προς τα εκεί, όχι κατά περίπτωση, εκ των υστέρων δηλαδή, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό έγινε, ε, πρέπει να είναι κομμάτι της πολιτικής συνοχής, αναπόσπαστο μέρος της. Και κλείνοντας, Είμαστε ε, ικανοποιημένοι από τη γενική κατεύθυνση που επέλεξε η Επιτροπή, αλλά πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην περιφερειοποίηση της πολιτικής, στα κοινωνικά ζητήματα και στο να καταστεί πιο πράσινη η πολιτική, κυρίως όσον αφορά τη διάσταση του κλίματος. Θα προτείνουμε τροπολογίες, κάποιες είναι ίσως λίγο τεχνικές, αλλά θα, δώσουν μια σοβαρή, θα προσφέρουν σοβαρή βελτίωση στον κανονισμό. Καθώς το συζητάμε σήμερα το θέμα, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε για την σημασία της πολιτικής συνοχής του ERDF και για τον προπολογισμών που πρέπει να προωθηθούν. Όλοι όμως αντιλαμβανόμαστε και την πίεση που υφίσταται ο προπολογισμό της Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ε, στις προτάσεις για τον προπολογισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα ε, όσοι συμμετάσχουν στον τριμερή διάλογο Εμεί, όπω ξέρετε, δεν, δεν συμμετέχουμε. Ελπίζω, λοιπόν, να, είναι... να πετύχουν όσοι θα υπερασπιστούν αυτή την πολιτική στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Δεν βλέπω τους άλλους ε, ε, συντονιστές της Επιτροπής ε, Ρέτζι. Θα δώσω, λοιπόν, το λόγο στον κύριο Φαν Μέστερόι να συνεχίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία σε αυτή τη φάση με την παρουσία της Επιτρόπου. Πολλά πράγματα υπόθηκαν θα ήθελα να πω ότι αν δει κανεί την πρόταση τη Κομισιόν, η πολιτική συνοχή εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα των στόχων και των δράσεων τη Ευρώπη. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν λιγότερα χρήματα ε, λόγω των αποτελεσμάτων και των νέων κρατών μελών είναι μια λογική συνέπεια όσο λυπηρό και αν είναι αυτό για τις δαπάνες, για τις υποδομές. Αυτό είναι το βασικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι η συνοχή θα πρέπει να παραμείνει σε αυτή τη θέση που έχει. Ε, όπως είπα προηγούμενος ομιλητής, αν πάρουμε την εσωτερική μετανάστευση, πραγματικά ε, περιμόνονται ε, κάποιες ε, περιοχές. Μέρη της ε, Πολωνίας, η Ρουμανία ε, Κάποιε περιοχές έχουν χάσει το μισό πληθυσμό του λόγω της γύρανση και λόγω του ότι ελκύεται ο πληθυσμός προς κάποια άλλα σημεία της Ευρώπη, σε κάποια κέντρα αριστεία και έτσι εγκαταλείπουν τα μέρη τους. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να δώσουμε μια απάντηση στους ανθρώπους σε αυτές τις περιοχές που καθυστερούν, που υστερούν στην ανάπτυξη. Σκεφτείτε ένα χωριό που έχουν φύγει όλοι οι νέοι, που μένουν μόνο οι γέροι. Και ε, τι να πούν αυτοί, ναι, πιστεύε, πιστεύουν στο ευρωπαϊκό project. Ε, η ερώτηση είναι τι έχετε υποσχεθεί, ε, ποιο ευρωπαϊκό έργο έχετε υποσχεθεί για τις δουλειές και για την ανάπτυξη. Ο, ε, νικητής τα παίρνει όλα. Ε, πρέπει να δώσουμε μία απάντηση ε, στο πρόβλημα αυτό μέσω της περιφερειακής πολιτικής. Το είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι ότι έχουμε κάποια μέσα στη διάθεση μας, κάποια εργαλεία. Έχουμε ακόμα μια αρκετά ισχυρή πολιτική συνοχή η οποία ευθυγραμμίζεται με άλλες πολιτικές. Είμαι εισηγητής ε, τώρα για το πρόγραμμα Horizon 2020. Ας είμαστε σαφείς, 90% των 120 δισεκατομμυρίων πάνε στα παλιά κράτη-μέλη. Εκεί είναι τα πιο καλά πανεπιστήμια. Εκεί, προς εκεί ε, έλκονται οι μεγαλύτερες επενδύσεις, προς τα εκεί. Πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο της γνώσης υπάρχει θεματική συγκέντρωση και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ας μην κοιτάξουμε το κάτω άκρο των επενδύσεών μας, αλλά και το άνω άκρο. Να δούμε πού μπορούμε να έχουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσω αυτής της συνεργασίας. Μιλάω για τις θεματικές συνεργασίες. Και μετά έχουμε αυτά τα νέα εργαλεία Ας δούμε την ε, καινοτομία για την, ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την καινοτομία και την ε, τεχνολογία. Υπάρχουν, ξεκίνησε πέρυσι, υπάρχουν 40 ε, σημεία όπου λειτουργεί αυτό το μέσο. Και πάλι είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι 80% είναι στα παλιά κράτη-μέλη, 10% στα νέα κράτη-μέλη. Άρα Όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση και την έξυπνη εξειδίκευση, υπάρχουν τόσο, τόσο πολλές δυνατότητες. Μιλάμε για την ενεργειακή μετάβαση, για τα νέα υλικά, για τη βιομάζα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία για την κλιματική αλλαγή επίσης. Τα πιο απόμακρα σημεία της Ευρώπης έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε μόλις η κυρία Κρέλ, ότι μέσω της πολιτικής συνοχής και του προϋπολογισμού μας πρέπει να βρούμε λύσεις και ευκαιρίες εξειδικευμένες για τα κράτη-μέλη και τις περιφερειές τους, όπου ένας να, να, να κάνει τρία, να επιτύχουμε ε, μεγαλύτερη ταχύτητα. Και αυτό ε, υπάρχει και στην πρόταση μου ότι η κάθε χώρα ε, σε επίπεδο περιφέρειας μπορεί να μεταφέρει 5% από τα ταμεία συνοχής σε project, παραδείγματο χαρή, που ανήκουν στην λογική του ορίζοντα 2020. Με άμεση μεταφορά, αφού ελεγχθούν εξονυχιστικά οι στόχοι και τα αποτελέσματα μέσω ε, αυτών που υπάρχουν στο φάκελο του κράτους μέλους. Αυτές είναι, αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τις μελλοντικές πολιτικές. Τώρα, για τα μικρότερα κονδύλια. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω εδώ. Πώς πρέπει να εξοδευτούν αυτά τα κονδύλια. καλύτερο τρόπος αξιοποίηση των κονδυλίων. Και ε, το θέμα των ε, μη δημόσιων επενδύσεων. Και επιπλέον, αν δούμε ότι κάθε ευρώ που βάζει η Γερμανία στην πολιτική συνοχή αποδίδει 1,5 ευρώ, από την εσωτερική αγορά γιατί παράγουν, εξάγουν και παίρνουν πίσω τα χρήματά τους. Από τις χρηματοοικονομικές αγορές επίσης, από την πραγματική οικονομία, από τα ευρωπαϊκά έργα. Για την Ολλανδία είναι 1,4 ευρώ πίσω που παίρνουν για κάθε ένα ευρώ. Άρα εδώ ε, πρόκειται για μια κεντρική πολιτική προς την οποία όχι κατακαιρματισμένη πολιτική προς την οποία πρέπει να κινηθούμε για να επιτύχουμε τους στόχους και τη συνοχή και όλους τους άλλους στόχους που έχουμε για τις γνώσεις, την ανταγωνιστικότητα, το κλίμα, ε, την πιο ε, πράσινη και έξυπνη Ευρώπη με ανάπτυξη και απασχόληση. Είναι σημαντικό λοιπόν η συζήτηση αυτή να γίνει εδώ όχι μόνο με τους φίλους μας της Επιτροπής Κότερ και στην Επιτροπή Ρέτζιερ αλλά γίνει μια πλήρη συζήτηση στην Ολομέλεια γιατί ε, έχουμε εκλογές, εμφανίζεται αυτό το κύμα του ε, αντιευρωπαϊσμού, του εθνικισμού, ε, πρέπει να στραφούμε στις περιφέρειες, όχι μόνο δίνοντας χρήματα, αλλά και με ένα νέο τρόπο επικοινωνίας. Σήμερα το βράδυ, ε, κυρία Επίτροπε, έχουμε ε, την απονομή των βραβείων ε, Regional Stars. Τώρα η συγγήτριά μας για την Ευρωπαϊκή ε, Εδαφική Συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ που επαναδιατυπώσατε την υποστήριξή σας στην, Επιτροπή, στην Πολιτική Συνοχή σε ένα πλαίσιο δημοσιομικό αρκετά ε, τεταμένο και σε ένα πολιτικό πλαίσιο αρκετά ανησυχητικό. Βέβαια, η πολιτική συνοχής αφορά την περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν τρεις πτυχές. Ε, ο κύριος Νίστερο είπε σωστά ότι πραγματικά πρόκειται για μια πολιτική συνοχή που δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει περισσότερη ανάπτυξη, λιγότερα ε, χάσματα στην Ευρώπη, οικονομικά, εδοφικά εδαφικά, να μην υπάρχουν σημεία ρήξης ε, κοινωνικά επίσης. Πολλοί ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη, και η κυρία Κρέλ ιδιαιτέρως, την ανάγκη να έχουμε μια πολιτική που να είναι πολιτική υπέρ των περιφερειών, ε, επαναδιατυπώνοντα βεβαίω και επιβεβαιώνοντα την αρχή τη επικουρικότητα. Και δεν πρόκειται για μια πολιτική των κρατών. Όσον αφορά την ομάδα μας, την Επιτροπή των Περιφερειών και την έκθεση που είχα αναλάβει κατά την περίοδο των διακοπών φέτος, ε, μιλάω για την έκθεση που αφορά την πρόταση της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ε, ακούγοντας όλους τους ομιλητές έχω την εντύπωση ότι εργαστήκαμε καλά παρά την πίεση που είχαμε από τις διάφορες προθεσμίες και παρόλο που θα υπάρχουν διαφορές βεβαίως και θα ε, υπάρχουν και τροπολογίες πολλές φορές ε, αντιφατικές, έχω την εντύπωση ότι ε, συγκλίνουμε σε κοινέ θέσεις πέρα από τις ε, πολιτικές μας πεπιθήσεις ο καθένας. Όσον αφορά την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, ε, η φυσικά εμείς ε, αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια κάποια συγκίνηση, κάποια ε, ε, ιδιαίτερα αισθήματα στις διάφορες περιφέρειες για τα θέματα αυτά. Ε, υπάρχει το πρόβλημα του προϋπολογισμού, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν εκεί. Ιδιαίτερα για, την, για τον τέταρτο πυλώνα που αφορά το Interreg και που ε, επηρεάζεται πάρα πολύ από το θέμα του προϋπολογισμού. Ένα άλλο που ενδιαφέρει όλους τους εμπλεκόμενους είναι η θαλάσσια συνεργασία τα είδαμε αυτά και σε όσα είπε ο κ. Ζουλό. Υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με αυτό το θέμα της ε, θαλάσσιας συνεργασίας που εντάσσεται σήμερα το πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας και στα διάφορα εδάφη, τα νησιωτικά όπως είναι η δική μου περιοχή, αλλά και στο Βορρά, στην Εσθονία συγκεκριμένα ε, και στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη Φιλανδία. Όταν είναι κανείς παράκτια περιοχή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σύνορα. Είτε είναι θαλάσσια σύνορα είτε χερσαία. Παραμένουν σύνορα. Και γι' αυτό ε, πολλοί εμπλεκόμενοι μα ζητούν να γίνει κάτι για το θέμα αυτό ε, και η θαλάσσια συνεργασία να παραμείνει στο πεδίο της διασυνοριακής συνεργασίας. Επίσης, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι ε, έχουν ένα αίτημα σχετικά με τα περίφημα 25 χιλιόμετρα που εισήχθησε και που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις. Σήμερα, για να μπορέσει να συνεργάζεται μια περιοχή με μια άλλη διασυνορική περιοχή, πρέπει πει ο πληθυσμός της κατά 50% να είναι εγκαταστημένος στα σύνορα, σε μια ε, απόσταση 25 χιλιόμετρων. Όταν βέβαια μιλάμε για ένα ορεινό σύνορο, δεν υπάρχει τόσο μεγάλος πληθυσμός από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, πολύ περισσότερη ανάγκη συνεργασίας στις περιπτώσεις αυτές ε, τους τελευταίους δύο μήνες συναντήθηκα με παραπάνω από 120 stakeholders, ενδιαφερόμενους φορείς και άκουσα όχι επικρίσεις αλλά άκουσα την βούληση να πούμε ότι ό,τι ε, αποδίδει θα πρέπει να διατηρηθεί. Ένα είναι αυτό και η βούληση επίσης εκφράστηκε να συνεχιστεί η συνεργασία. Και αυτό εξίσου σημαντικό είναι στα σημερινά πλαίσια και στο σημερινό κλίμα. Με τη συνάντηση με τον κύριο Άρημον, ε, ε, είδα ότι επίσης ε, συμφωνούμε στα περισσότερα σημεία Επίσης με την κυρία Μαρίνη και τον κύριο Σνάιντερ, ε, οι συναντήσεις αυτές έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία σαν ένας σημαντικός άξονας συνοχής. Για τα δύο-τρία σημεία που θα ήθελα ιδιαίτερως να υπογραμμίσω, είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκφράσουμε την ε, ικανοποίησή μας Υπόθηκε αυτό, αλλά γιατί να μην το ξαναπούμε αφού είναι κάτι θετικό. Η αρχή, για την αρχή της ε, απλούστευσης, για την εδαφική συνεργασία, είτε πρόκειται για τις βασικές αρχές της απλούστευσης, είτε για το να το υπόψη τα μικρά έργα ε, εδαφικής συνεργασίας, είτε πρόκειται για τις μακροπεριφέρειες είτε πρόκειται για την ανάγκη να καθοριστούν καλύτερα οι θαλάσσιες λεκάνες. Όλα αυτά τα σημεία ε, έγιναν δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σημείο όπου γίνονται ακόμα συζητήσεις και σίγουρα θα γίνουν και στο μέλλον και στην Επιτροπή μας και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Κοτέρ αλλά πολύ ε, σίγουρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για την, ε, το τέταρτο πυλώνα, το, το Interreg συγκεκριμένα, όπου υπάρχει η, ε, σαφώς το αίτημα να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός και, μετά στον πυλώνα 5 της ε, εδαφικής συνεργασίας που πρόκειται για μια καινοτομία καθ' αυτή, δηλαδή μια πρωτοβουλία υπέρ των διαπεριφερειακών επενδύσεων για θέματα καινοτομίας. Από τη μία πλευρά θεωρούμε ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Όπως είπε και η κυρία Επίτροπος προηγουμένως, ναι, η καινοτομία είναι απαραίτητη στις περιφέρειες και ναι, επίσης είναι απαραίτητο οι περιφέρειες να συνεργάζονται ε, στον τομέα των επενδύσεων για την καινοτομία, για την ε, προηγμένη τεχνολογία, για να έχουμε το αποτέλεσμα της αλλά φυσικά αυτό δεν πρέπει να περιορίζεται στις λίγες πιο ανταγωνιστικές, ε, πιο αποδοτικές ε, περιφέρειες. Όπως είπαν πολλοί ομιλητές, πραγματικά σήμερα ε, θεωρούμε κάτι το αυτονόητο, σαν αυτονόητο μάλλον, ότι ε, οι ε, επιδοτήσεις για την καινοτομία και τις επιδόσεις πάνε στις περιφέρειες που ήδη είναι οι πιο καινοτόμες και έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Ε, υπογραμμίζουμε λοιπόν ακόμα μια φορά το απαραίτητο. Ε, είναι αναγκαίο ε, τα μέσα αυτά να είναι ανοιχτά για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Όχι μόνο για αυτές που είναι ήδη πολύ προχωρημένες, σούπερ ανταγωνιστικές, ε, ε, ε, που έχουν όμως ε, αλλά και σε αυτές που έχουν κάποια διαρθρωτικά προβλήματα αλλά μπορούν να καινοτομήσουν, μπορούν να προσφέρουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η μελλοντική πολιτική της εδαφικής συνεργασίας που θέλει να είναι καινοτόμος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις περιφέρειες και για τον πυλώνα 5. Και για να κλείσω, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, το είπαν εξάλλου αυτό και άλλοι ομιλητές, να διατηρήσουμε την κλίμακα των περιφερειών σαν την ε, σωστή κλίμακα, το σωστό επίπεδο όπου μπορεί να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όσον αφορά την πολιτική συνοχή και εδαφική συνεργασία. Ε, είναι πάρα πολύ γνωστή η διάσταση αυτή. Το Interreg θα έλεγα σήμερα ότι είναι το πιο αναγνωρίσιμο πρόγραμμα στην Ευρώπη μαζί με το Erasmus. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συνοχή, πρέπει να τη διατηρήσουμε ε, στο σημερινό πολιτικό ε, ε, περιβάλλον το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλες ε, ε, αβεβαιότητες σε κάποιες χώρες και θα πρέπει να διατηρήσουμε ό,τι πάει καλά, ό,τι αποδίδει. είτε σε διασυνοριακό επίπεδο είτε σε άλλο επίπεδο να, ε, να διατηρήσουμε τις καλές αυτές περιπτώσεις που έδωσαν τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες τα τελευταία αυτά χρόνια να οικοδομήσουν έργα αποδοτικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε. Θα μιλήσω ρουμάνικα. Και θα είμαι σύντομος. Έχουμε δύο περιορισμούς που τους έχουν υπογραμμίσει πολλοί ομίλητες και θα τονίσω εγώ κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Είμαστε όλο τόσο ε, σύμφωνοι μεταξύ μας που μοιάζει να έχουμε αφήσει τις ιδεολογίες μας ε, στην είσοδο για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα της πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Επίσης, πρέπει ο στρατηγικός προσανατολισμός του νέου αυτού προγράμματος πραγματικά να εξυπηρετεί τις ανάγκες ε, της οικονομικής και ενεργειακής μετάβασης. Ο συνάδελφος Μίλτενμπουργκ ανέφερε ότι πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό για την έκθεση του IPCC του Διεθνούς Οργανισμού για την Κλιματική Αλλαγή. Ο τίτλος του ήταν «Ξυπνήστε ηλίθιοι». Δημοσιεύτηκε χθε. Αυτό είναι το μήνυμα που απευθύνεται προς ε, αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εάν δεν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε μέσω της πολιτικής συνοχής, μέσω και του InvestEU και όλα τα άλλα μέσα για να, για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει τον πρωτοπόρο της ρόλο σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και χορήγησης οικονομικής βοήθειας προς τις χώρες που έχουν πολλές προκλήσεις κλιματικής αλλαγής. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, τότε τα λόγια θα μείνουν λόγια. Τα λόγια που είπαμε και για να ληφθεί η απόφαση των Παρισίων και αυτά που θα πούμε εν ώψη της περίοδου. Η απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι τεράστια. Αυτά που αναφέρει η έκθεση του IPCC λένε ότι μέχρι το 2050 η κατάσταση θα έχει γίνει αφόρητη αν υπάρξει αύξηση άνω του 1,5 βαθμού. Και αν η αύξηση αυτή είναι 2 βαθμοί Κελσίου, τότε η κατάσταση θα είναι τραγική. Τώρα σε επανέλθω σε πολύ πιο απτά θέματα. Συμφωνώ με τις θετικές επιπτώσεις των αποφάσεών μας εν ώψη των ευρωεκλογών. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι θα εκλεγούν για το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εκλεγούν ε, υποστηρικτές ή αντίπαλοι της Ευρώπης. Γιατί εάν επικρατήσουν ε, οι μεν, ε, θα είναι πολύ διαφορετική εξέλιξη της Ευρώπης από ό,τι αν επικρατήσουν οι δε. Και η πολιτική συνοχή πρέπει να είναι ε, το μεγαλύτερο όπλο μας για να επιδιωχθεί το σωστό αποτέλεσμα. Κυρία Επίτροπε, το θέμα δεν είναι να υπάρξουν ε, δραματικές αλλαγές στην ισχύουσα πολιτική, διότι οι διαχειριστικές αρχές, οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές τώρα γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά και θα μπορέσουν να τα εφαρμόσουν ταχύτερα εάν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές οι οποίες θα επιβραδύνουν την εφαρμογή και επίσης θα έχουμε και τις επιπλοκές που θα προκύψουν και πάλι εάν επαναληφθεί η καθυστέρηση που υπήρξε το 2014 για την έγκριση των νομοθετημάτων και των ε, χρηματοδοτήσεων. Οποιαδήποτε αιρεσιμότητα, είτε είναι οικονομική αιρεσιμότητα, είτε πολιτική αιρεσιμότητα, με τη γενικότερη ένα του όρου θα βλάψουν την έκφραση αλληλεγγύης και αυτό όχι στο μέλλον αλλά τώρα ε, εν ώψη των ευρωεκλογών επίσης ξέρετε ότι ε, σε πολλά κράτη-μέλη οι αντιλήψεις αυτές για Ευρώπη πολλών ταχυτήτων ή ε, ομόκεντρο κύκλων θεωρούνται ως ε, προσπάθεια για να διατηρηθούν οι διαφορές ανάπτυξης ε, μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και άρα ως μια προσπάθεια κατά της εξέλιξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό που ανέφεραν και άλλοι ομιλητές Δηλαδή ότι πρέπει να διατηρηθεί το 1 3. Γιατί υπάρχουν ε, πολύ μεγάλες ε, διαφορές επίπεδου μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού. Είναι αδιανόητο ότι η πρώτη πρώτου του 2021 να είναι έτοιμα, έτοιμα όλα τα ε, εφαρμοστικά μέτρα και μηχανισμοί. Οι περιφέρειές μας δεν θα είναι σε θέση να απορροφήσουν τους πόρους αν γίνει κάτι τέτοιο. Να μην έχουμε αυταπάτες περί αυτού. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί βέβαια ένα κριτήριο επιλεξιμότητας για το Ταμείο συνοχή. Όπως συνεργάζομαι με τον συνάδελφο Κοτσολίν. Πρέπει να διατηρηθούν ως επιλέξιμα τα προγράμματα που αναφέρονται στο τροχαίο υλικό. Γιατί ξέρετε ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ε, ή λιγότερο ρηπαίνουσε. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τη χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων. Ε, να μην ξεχνάμε ότι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ο χειμώνα διαρκεί πάρα πολύ. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να γίνει ενεργειακή μετάβαση. Γι' αυτό πρέπει να μπορούμε να έχουμε δίκτυα περιφερειακής ε, ε, θέρμανσης. Έτσι θα δώσουμε μια ευκαιρία στις χώρες αυτές να μην επενδύσουν στον άνθρακα αλλά στο φυσικό αέριο. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι πόροι για αυτές τις ε, περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούν να γίνει η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι δυνατόν να τους υποσχόμεθα ότι τα ωφέλη θα τα έχουν ε, στην μεταθανάτιο ζωή γιατί μόνο η βίβλος ε, εγγυάται την ε, ζωή μετά θάνατον. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ε, ελλειπούς απορρόφησης των πόρων. Και κάτι ακόμη για το ΣΕΦ. Κυρία Επίτροπε, το Ταμείο Συνοχής προβλέπει 10 δις για το ΣΕΦ, τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό είναι ουσιώδες. Πρέπει να διδρυθούν οι κανόνες για τρία χρόνια, κατά τα οποία πρέπει να διατηρούνται ε, ως εθνικοί πόροι οι πόροι που έχουν ε, αποδοθεί και μόνο μετά να περνάνε στο γενικότερο πλαίσιο. Να μείνουν οι ίδιες οι προδιαγραφές. Έτσι θα έχουμε λιγότερη ε, αντίδραση και είναι σημαντικό οι κανόνες για τις μεταφορές. Να αναφέρονται στο γενικό κανονισμό. Όσον αφορά ε, τους ε, κανόνες για το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Αυτός ο κανόνας για τα μεταφορέ πρέπει λοιπόν να αναφέρεται μόνο στο γενικό κανονισμό αλλά και στους επιμέρους κανονισμού για τα ταμεία και για το συνδέοντα στην Ευρώπη. Και κάτι ακόμη. Το συνδέοντα στην Ευρώπη λένε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και ω πλατφόρμα για τη στρατιωτική κινητικότητα που θα χρηματοδοτείται βέβαια από τους αμυντικούς προπολογισμού. Αλλά πρέπει να έχουμε κανόνες για να υπάρχει συμβατότητα. Γιατί αλλιώς θα βασίζεται και στην ε, προσέγγιση συνοχής και στην αμυντική ε, προοπτική και στην ε, προοπτική της στρατιωτικής κινητικότητας. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συντονισμός μεταξύ της δράσης της ε, υπηρεσίες εξωτερική δράση με την ε, πολιτική ε, για την κινητικότητα. Ο κύριο Σάντσο Μουνιώθ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την εισηγήτρια τη έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την πρόεδρο Σουζάνα Ντίαθ της τοπική κυβέρνηση Ανδαλουσίας. Και θα ασχοληθώ λοιπόν με τις ε, διαβουλεύσεις που κάναμε με τους κοινωνικούς εταίρους και θέλουμε να τονίσουμε ορισμένα θέματα για το κοινωνικό ταμείο. Το πρώτο είναι, είναι ότι θέλουμε να συνδεθεί καλύτερα η πρόταση κανονισμού με τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύνοχης, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να μην είναι απλώς ένα όργανο κοινωνικής πολιτικής, Κατηγορηματικά απορρίπτουμε την ε, πολύ περιορισμένη παρουσία και ορατότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών που προβλέπονται. Πρέπει να αναφερθεί ο ρόλος που παίζουν, γιατί έχουν πολύ ευρεία ε, εμπειρία βεβαίως. Επίσης θέλουμε έναν προπολογισμό που να είναι επαρκής για το Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ γιατί πρέπει να ασχοληθεί και με άλλα θέματα όπως η υγεία, η κατάρτιση και η κατάρτιση συγκεκριμένα των ε, μεταναστών. Βεβαίως πρέπει να συντονίσει τις ενεργειές του Ταμείου αυτό με το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Θα συζητήσει η Ολομέλεια της Επιτροπής μας την έκθεση αυτή το απόγευμα. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μετανάστες. Στην Ανταλουσία, όπως θα ξέρετε, η ακτή μας ε, απέχει 14 χιλιόμετρα την Αφρική. Ε, δεχόμαστε κύματα μετανάστευσης και ιδιαίτερα ε, ευάλωτα άτομα, ασυνόδευτα, ασυνόδευτα ανήλικα άτομα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να τους παράσχουμε ως μέσα υπηρεσίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συντονισμός και της επιγούσης βοήθειας και της κατάρτισης και εκπαίδευσης για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Στηρίζουμε επίσης αυτό που υπόθηκε για την περιφερειακή συνεργασία. Μα είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η κυρία Κρέτου είπε ότι είναι σημαντική επιτυχία είναι μια σημαντική επιτυχία το Εράσμους και έχουν ε, σημειωθεί πολλά πράγματα λόγω αυτού. Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να αποτελέσει το εράσμους των περιφερειακών αρχών. Μπορεί ε, να γίνει αυτό στη θάλασσα ή και αλλού. Υπάρχει όμως αληθινά σύγχυση στον τομέα της θαλάσσιας συνεργασίας. Η δική μου περιφέρεια έχει εδαφική και ε, συνεργασία στην Ξηρά με την Αλγκάρβ. Αλλά έχουμε και θαλάσσια συνεργασία με το Μαρόκο, το οποίο πρέπει να συμπεριλάβουμε στον τομέα της μετανάστευσης και σε άλλους τομείς. Όμως, για, όσον αφορά τη θαλάσσια συνεργασία, υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει στενός δεσμός. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει σύραγγα και παρόλα αυτά συνεργαζόμαστε επί 25 χρόνια. Τα όρια της Ανταλουσίας δεν είναι απλώς ε, ισπανικά όρια σύνορα, είναι ευρωπαϊκά. Και επίσης πρέπει να συνδυαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα για να μειωθούν οι κοινωνικές ε, ανισότητες και να επενδύσουμε στα άτομα, στους πολίτες που έχουν δει περισσότερο από την κρίση. Έτσι θα αντιληφθεί καλύτερα η κοινή γνώμη, το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ίσως ε, να απομακρυνόμεθα από την κρίση, αλλά δεν θα λήξει η κρίση παρά μόνο όταν βοηθήσουμε τους πάντες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν να βραδιπορεί γιατί έτσι θα αγγιθούμε και το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία... Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μαλέτιτς. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και λίγο χρόνο στην κυρία Πίτροπο. Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω με την ε, Επιτροπή των Περιφερειών επί του πολύ σημαντικού αυτού θέματος. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε υποστηρικτές πολιτικής συνοχής και παλεύουμε για την, ε, να είναι ισχυρή η πολιτική αυτή και τώρα πραγματικά πρέπει να πολεμήσουμε, να παλέψουμε με βάση όσα έχουμε το, θέμα μετά την πρόταση της Επιτροπής ε, είναι θέμα αν θα παραμείνει ισχυρή ή όχι γιατί όπως ε, κάποιοι από εσά ήδη είπατε έχουμε σοβαρές περικοπές στο πλαίσιο του ε, δημοσιονομικού πλαισίου για την ε, πολιτική συνοχής ε, περικόπτεται κατά 10% η πολιτική συνοχή, ενώ ταυτόχρονα ε, αυξάνονται κατά 50% ή και 100% κάποια προγράμματα ανταγωνιστικότητα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό που λέμε όμω είναι ότι προσφέρουμε ε, περισσότερε δυνατότητε στι πιο ανταγωνιστικέ περιφέρειε και λιγότερε δυνατότητε και ευκαιρίε στι λιγότερο ανταγωνιστικέ περιοχέ. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό και θα ε, προετοιμάσουμε μια άλλη πρόταση. Κάτι άλλο που κάποιοι προλύσαντες ανέφεραν ε, είναι αυτό που έχει σχέση με το Ταμείο Συνοχής. Η περικοπή του Ταμείου Συνοχής κατά 46% τι συνεπάγεται. Ε, είναι ένα μέσο που χρειαζόμαστε. Αν έχουμε μόνο τους μισούς πόρους, τι σκοπεύουμε να κάνουμε, ποιος είναι ο στόχος μας. Είναι σαν να μην το θέλουμε πια. Αν δεν το θέλουμε ε, στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής, ενώ είναι από τα βασικά μέσα. Το ερώτημα λοιπόν και πάλι τίθεται, τι θέλουμε να πετύχουμε και πέραν όλων αυτών ε, επιτρέπουμε την εύκολη μεταβίβαση των ε, το, της ε, πολιτικής συνοχής προς άλλους τομείς. Γιατί να μην συμβαίνει το αντίστροφο, να ε, προστίθενται στην, στην πολιτική συνοχή αλλά μέσα. Ε, γιατί πλέον ε, με τη θέλησή τους τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συνεισφέρουν μέχρι και 5% ε, κάθε ταμείου προς το νέο μέσο. Και αυτό είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί αυτό το νέο μέσο επενδύσεων και θα υπάρχει ο πειρασμός να γίνει αυτό. Επίσης αυτή η μεταφορά των 10 δισεκατομμυρίων του ε, μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Αφού το Ταμείο έχει ήδη μειωθεί κατά 46%. Τελικά ποιο είναι το μέλλον τη πολιτική συνοχής. Επίση, θέλω να αναφέρω ότι αυτέ οι μακροοικονομικέ αιρεσιμότητε που ισχύουν και ε, υπάρχει και η πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων, του οποίου προϋπολογισμός είναι 25 δις ευρώ. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε στον κανονισμό μας, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, να έχουμε το αίτημα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα τους πόρους της πολιτικής συνοχής για την στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Γιατί, αφού υπάρχει ένα νέο ε, ταμείο των 25 δις και παρόλα αυτά αυτό πρέπει να συμπληρωθούν τα 25 εκατομμύρια από την περιοχή, από την ε, πολιτική συνοχής. Γιατί όχι να μην κάνουν το αντίστροφο. Πρέπει να το αρνηθούμε αυτό. Ε, είναι σημαντικό. Η πρόταση όμως της Κομισιόν δεν στηρίζει την πολιτική συνοχή παρά την περικόπτη και την σταματά. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό. Και ακόμα κάτι. Στο νέο κανονισμό υπάρχουν πολλοί όροι και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Στον τρέχοντα κανονισμό ξεκινήσαμε με, από την τρέχουσα περίοδο με τις ερεσιμότητες και τις εκ των προτέρων και την εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Τώρα στο νέο κανονισμό επιπλέον έχει βελτιωθεί η εξάντε ερεσιμότητα αλλά έχουμε ερεσιμότητα παραβίασης που επανεισέρχεται και το θέμα του κράτους δικαίου. Δηλαδή κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η πολιτική συνοχή να γίνει πιο σύνθετη και να σταματήσουμε τα, τα, τους πόρους του Ταμείου Συνοχής να φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. λόγω της κακής διακυβέρνησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι θετικό. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής ε, από την Επιτροπή των Περιφερειών από το ECR. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Θα είμαι σύντομο, Πολλά από όσα είπα, από όσα ακούστηκαν, ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Ε, το θέμα τη συνεργασία την παρακολουθώ ε, από τα τελευταία χρόνια και είμαι και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Περιφερειών. δύο πράγματα για τον προπολογισμό τη διαμεθοριακή συνεργασία. Μιλήσαμε για το μέλλον τη πολιτική συνοχή και του προπολογισμού. Πάντοτε αναφερόταν το θέμα τη προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η κατευθυντήρια αρχή μας. Δεν ξέρω καλύτερο τέτοιο παράδειγμα από ότι η διαμεθοριακή συνεργασία. Έγινε και η διάσκεψη με την κυρία Μιχαήλοβα εδώ το Μάρτιο και υπήρχε μεγάλη συνένεση. Συμμετείχατε κι εσεί. Η διαμεθοριακή συνεργασία ε, συμφωνήθηκε, πρέπει να στηριχθεί και να αυξηθεί σημαντικά. Δυστυχώ οι προτάσει δεν το ε, δείχνουν αυτό. Ε, μιλήσαμε για 6,5 δις αύξηση ε, στην κινητικότητα. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από ότι το σύνολο της ε, διαμεθοριακής συνεργασίας ε, για τους πολίτες. Και διαρωτώμεθα, ε, μήπως θα πρέπει τα χρήματα να πάνε κάπου αλλού, τα ξοδεύουμε σωστά. Αλλά η συνεργασία δεν είναι μόνο χρήματα, χρειάζεται και το περιβάλλον. Θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν για την αναθεώρηση του, του διαμεθοριακού σκέλους και τις προτάσεις για τον διαμεθοριακό μηχανισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή βελτίωση. δεν μας απασχολεί μόνο το Interreg, αλλά και το θέμα πέρα από αυτό. Το θέμα επίσης της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους, πολιτικέ, με τους πολίτες μέσω της πολιτικής ε, ε, συνοχής. Εγώ ζω στο, στα σύνορα της Τσεχίας, Πολωνίας, Γερμανίας. Έχουμε 2.000 συμμετέχοντες στα έργα που, στις εκδηλώσεις που οργανώνται λόγω του Ίντρεγκ. Και πολλά από αυτά είναι μικρά έργα. Υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Έγινε μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Ε, για πρώτη φορά ε, φέραμε το το Ταμείο για τα Μικρά Έργα στον κανονισμό NDC και μπορέσαμε να τον παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Ρέτζιο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα ε, προς την ε, πολιτική συνοχής της διαμεθοριακής συνεργασίας ε, στα μάτια των πολιτών. Και τέλος ένα σημείο όσον αφορά την απλούστευση. Είναι μεγάλο το θέμα του αριθμού των ελέγχου Θα αναφερθώ και πάλι όμως μόνο στη διαμεθοριακή συνεργασία η Κομισιόν προτείνει για μικρά έργα κάτω των 100.000 ευρώ η απλουστευμένη επιλογή κόστους θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Αυτό αφορά το πρόγραμμα. Εγώ είμαι ο δικαιούχος, ε, χρησιμοποιώ κατά αποκοπήν ποσά ε, αλλά έχω και συγχρηματοδότηση από το δημοτικό ή κρατικό προπολογισμό. Μπορεί λοιπόν να έρθει ο εθνικό έλεγχος και να μου ζητήσει κάθε τιμολόγιο, να δικαιολογήσω κάθε ε, λεπτό που έχω ξοδέψει. Πρέπει να υπάρχει κάποια συμφωνία εδώ, κάποια εταιρική σχέση, ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που, στα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να ε, κυριαρχεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και έτσι να Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή εκ μέρου της Επιτροπής Ρέτζο, ο κύριο Ζουλό. Θα ήθελα να είστε σύντομο για να μπορέσει να απαντήσει η επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Να υπενθυμίσω ότι πολλοί είπαν ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ε, για να δούμε αυτές τις προτάσεις που διατυπώθηκαν. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ και λίγους μήνες δεν είμαστε βέβαιοι ότι καν θα υπάρχει πολιτική συνοχή ε, η οποία θα ωφελήσει το σύνολο των ε, περιφερειών της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν τις προτάσεις που έχουμε τώρα ενώπιόν μας, τις συγκρίνουμε με τα νούμερα της προηγούμενης περίοδου. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή και είναι λογικό να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί, να κινηθεί η Επιτροπή Συνοχή, Πολιτική Συνοχής γιατί ε, βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο εδώ και 7 χρόνια. Η έβδομη έκθεση συνοχής, η οποία δημοσιεύτηκε από την Κομισιόν, δείχνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Φερρυπίν ότι σχετικά με την εξέλιξη αυτή κάποιες περιφέρειες γνώρισαν στην περίοδο αυτή σημαντική ε, ανάπτυξη, μερικές πολύ σημαντική, ενώ κάποιες άλλες ε, περιφέρειες ε, ε, αντιμετώπισαν ε, δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες από την κρίση. Επίσης, επισημαίνεται ιδιαίτερα η κατάσταση περιφερειών που έχουν μέσο εισόδημα, μέσα έσοδα και βλέπουμε ότι για αυτές υπάρχει κίνδυνος μείωσης αν δεν ε, ε, προσέξουμε επαρκώς την κατάστασή τους και ότι η σχέση, ε, η έκθεση έδειχνε ότι οι περιφέρειες που έχουν, αυτές είναι οι περιφέρειες με την μικρότερη ανάπτυξη. Αλλά πρέπει η Κομισιόν να διευρύνει την περίμετρο των περιφερειών που είναι σε μετάβαση, σε περίοδο μετάβασης αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε η Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Να περάσουμε ε, στο 70% για τη συγχρηματοδότηση των ε, περιφερειών που είναι σε μετάβαση. Και εν κατακλείδη, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων ετών χωρίς να αναφερθούμε στο Brexit. Γνωρίζουμε ότι πολλές περιφέρειες θα επηρεαστούν και μάλιστα έντονα και σκληρά από τις επιπτώσεις που θα ξεκινήσουν ε, ταχαίως από εδώ και πέρα όσον αφορά τη συνεργασία αλλά και τις ανταλλαγές οικονομικές, το εμπόριο, τις, περιφέρει, τις ε, μεταφορές και άλλους τομείς. Άρα ε, ήδη έχω πει ότι η Ευρώπη πρέπει να προβλέψει κάποιο ταμείο ή κάποιο ειδικό μέσο, κάποιο μηχανισμό εν πάση περιπτώσει για την προετοιμασία των περιφερειών κυρίως δε των περιφερειών που θα γίνουν ξαφνικά μεθοριακές, παραμεθόριες. Ε, ε, θα ήθελα λοιπόν, κυρία Επίτροπε, να ακούσω τι έχετε να πείτε από αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, έχετε τον λόγο για να προσπαθήσετε να απαντήσετε στα ερωτήματα. Βεβαίω ξέρουμε πάντα ότι ποτέ δεν αρκεί ο χρόνος για τις συνεδριάσεις μας. Έχετε τον λόγο. For me. Ευχαριστώ πολύ. Για μένα, όπως είπα, είναι πάντοτε χαρά και σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Βέβαια για κάποια θέματα δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις, αλλά συνολικά πιστεύω ότι η σημερινή συνάντηση είναι μια ακόμα επιβεβαίωση του, της κοινή μας κατανόησης για αυτή τη τόσο σημαντική ε, πολιτική και το μέλλον της, για το όφελος των πολιτών μας. Ο κύριος ε, Μποσνάρου, αρχίζει είναι συμπατριώτης μου και ξεκινάω με αυτόν και με όσα είπε, για μένα η πολιτική συνοχή δεν έχει πολιτικό χρώμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αφήσουμε πίσω όλες τις προκαταλήψεις μας και να περασπιστούμε αυτό το τόσο σημαντικό εργαλείο που είναι τόσο σημαντικό για όλες τις περιφέρειες. Λοιπόν, όλοι συμφωνούμε ότι όσον αφορά τη σημασία και τη σπουδαιότητα της πολιτικής συνοχής και ότι χρειάζεται συντονισμός ανάμεσα στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό ε, επίπεδο και γι' αυτό Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα βρίσκομαι όχι μόνο μεταξύ των ε, ε, αξιότιμων κυρίων Ευρωβουλευτών, με τους οποίους ε, συναντιέμαι συχνά, αλλά και με τους εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών. Γιατί εσείς τελικά είστε ο σύνδεσμός μας με τους πολίτες και ως εκπρόσωποι των τοπικών αρχών αλλά και των ψηφοφόρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποια σχόλια για το νομοθετικό πακέτο. Ξέρετε πολύ καλά ότι παρουσιάσαμε την πρότασή μας τον περασμένο Μάιο και φυσικά άκουσα προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια και τις ιδέες σας. Τώρα περιμένουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσάς δηλαδή, και από το Συμβούλιο να καταλήξουν στη θέση τους ο καθένας για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η σκέψη μου είναι να σας προκαλέσω να έχετε ένα φιλόδοξο σχέδιο ώστε να αρχίσει ο τριμερής διάλογος ε, τον Δεκέμβριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απευθύνουμε σε εσά, κυρία Πρόεδρε, ε, για να μην έχουμε καθυστερήσεις. Αν πραγματικά θέλουμε να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε γέρο τη νέα προγραμματική περίοδο, πιστεύω ότι πραγματικά η τελευταία μας ευκαιρία είναι να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο τον ε, Δεκέμβριο και το Μάρτιο επί Ρουμανικής Προεδρίας να έχουμε τη συμφωνία. Ε, όσο ανεξάρτητα από το πόσες γνώσεις έχει κανείς ή πόση μεγάλη πείρα ε, είναι σαφές ότι το νέο κοινοβουλίο δεν θα μπορέσει αμέσως να ασχοληθεί με τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να πραγματοποιηθεί πρόοδος σε αυτό το κοινοβούλιο. Ε, και όσο αφορά τους εκπροσώπους του Συμβουλίου ε, οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων ε, θα πρέπει να έχουν επίγνωση του τι σημαίνει μια καθυστέρηση για την πρόταση αυτή ε, πέραν των ε, ευρωπαϊκών εκλογών. Γιατί ε, πραγματικά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ούτως ή άλλως θα χρειαστεί χρόνος για να οργανωθεί εσωτερικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άρα θα έχουμε καθυστέρηση τουλάχιστον μισού έτους, ε, μισό έτο, το οποίο θα μας κοστίσει πάρα πολύ σε χρήματα που θα πρέπει να διατεθούν από το... Ε, τον εθνικό προπολογισμό και όχι ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα, όλες οι οικονομικές πτυχές της πρότασης αυτής θα συζητηθούν και θα επιληθούν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών που εκπροσωπούν τις χώρες τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά οι επιμέρους, κανονισμοί βρίσκονται στα χέρια σας, στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν σε λεπτομερή ζητήματα που τελικά βρίσκονται στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Σνάιντερ, ας πούμε, μίλησε για δείκτες για Ανατολική και Δυτική Γερμανία. Ε, η Ανατολική Γερμανία είναι φτωχότερη από την Δυτική Γερμανία όσο πιο πλούσια είναι μια περιοχή, τόσο λιγότερα χρήματα παίρνει. Αυτό είναι ο κανόνας. Τώρα, πώς θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα είναι θέμα των εθνικών και των περιφερειακών προγραμμάτων. Πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα προγράμματα αυτά από σήμερα ήδη, από αυτή τη στιγμή, κατά την τρέχουσα περίοδο και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να επιστρέψουμε στις χώρες μας, να συνομιλήσουμε με τις περιφέρειες και τις εθνικές κυβερνήσεις ούτω ώστε να αρχίσει να ε, ολοκληρώνεται αυτή η προγραμματική περίοδο ε, γέρο και να υπάρξουν και όριμα προγράμματα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Συμφωνώ με όλους σχεδόν για τη στρατηγική συμμαχία που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στην Επιτροπή των Περιφερειών, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και συμφωνώ και με το Συμβούλιο επίσης. Μια άλλη πρόταση για το εν διατονή συν υποβάλαμε την πρότασή μας με τον ίσιν 2 και με τις απαραίτητες εξηγήσει από τη μεριά μας αλλά τώρα ε, βρίσκεται πάλι στα δικά σας χέρια και η πρόταση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που είπε η Κωνσταντζέ η κυρία Κρέλ, είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται για business as usual. Είναι μια τεράστια ευθύνη που έχουμε μπροστά μας, ίσως και απέναντι στις ε, μελλοντικέ γενιές. Να βρεθούμε πιο κοντά στους πολίτες και να είμαστε σε θέση να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να αναχαιτήσουμε αυτό το ευρωσκεπτικιστικό ε, ρεύμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να το αποδείξουμε αυτό. Και βεβαίω καταλαβαίνω πολύ καλά ότι πρέπει να κάνουμε αμοιβέ προσπάθειε. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι σε χώρες όπου δεν επισκέφτομαι αυτοπροσώπω, τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν αναφέρονται καν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε παρόντες, όχι μόνο όταν εγκαινιάζεται ένα έργο, είναι ε, πια ε, στιγμή να σταματήσει αυτό το παιχνίδι. ότι όλα τα κακά προέρχονται από τις Βρυξέλλες και να ε, μην αναφέρονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτό είναι ε, δυστυχώς κάτι που συμβαίνει και σε επίπεδο περιφερειών αλλά και σε επίπεδο υπουργών. Ε, που έρχονται στα Συμβούλια Υπουργών και λένε ότι η έλλειψη επικοινωνίας ε, είναι το πρόβλημα μας, αλλά μετά γυρίζουν στις χώρες τους και εγκαινιάζουν ένα έργο χωρίς να αναφέρουν καν ότι έγινε με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, με ευρωπαϊκά ε, κονδύλια. Κάτι άλλο που έγινε πολύ σαφέ για μένα, το πρόγραμμα διασυνορικής συνεργασίας Interreg. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μια ανακοίνωση και Προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς θα τη μεταφράσουμε την ανακοίνωση αυτή στην πραγματικότητα. Εργαζόμαστε με ε, κατευθυντήριες γραμμές, ε, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ε, οργανώσουν σε εθελοντική βάση την διασυνοριακή συνεργασία. Ε, μια χώρα δηλαδή να χρησιμοποιήσει πιο προχωρημένη νομοθεσία που έχει το γειτονικό κράτος για μένα η διασυνοριακή συνεργασία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Μερικές φορές θεωρείται σαν κάτι δεδομένο γιατί όχι μόνο ε, οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά έχει και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι απουλώνει τις πληγές που υπάρχουν στην ε, Ήπειρό μας. Σλοβακία και Τσεχία, παραδείγματο χάρη, αλλά κάτω Αυστρία, και Βρατισλάβα, όπου πολλοί άνθρωποι ε, έχασαν τη ζωή τους και άλλα παραδείγματα όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παραμεθόριες περιοχές και τώρα ε, αναπτύσσονται μαζί, συνεργάζονται, έχουν πανεπιστήμια. Είναι αυτή η αντίληψη που έχουμε για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν, εφαρμο... δεν έγινε βέβαια στο Δουβλίνο ή στο Λονδίνο, δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες ε, και βοήθησε πάρα πολύ αυτές τις τόσο ε, ε ταραχώδεις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να έχει λοιπόν τη θέση του για μετά το 2020 και για την πολιτική ε, για το Brexit, συγγνώμη, αυτό μας επηρεάζει όλους, γιατί χάνουμε ένα καθαρό ε, συνεισφορία στον προϋπολογισμό της κοινότητας. Ε, θα δούμε ο, ο κύριος Μπαρνιέ τι έχει ε, επιτύχει στις διαπραγματεύσεις, ο οποίος υπήρξε και επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική στο παρελθόν και ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί μια οικονομική ρύθμιση και ξέρουμε ότι μέχρι το 2023 το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβάλει ό,τι οφείλει προς όλα τα κράτη-μέλη. Και βέβαια, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, δεν έχουμε αρκετό χρόνο αυτή τη στιγμή αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ήμουν στην, ε, συμμετείχα στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ε, Περιφερειών και πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. 6.000 άνθρωποι ήρθαν ε, στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα για να μιλήσουν και να συζητήσουν για την πολιτική συνοχής και δημοσιογράφοι κλπ. Και ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της εβδομάδας των περιφερειών ήταν ότι είχαμε πάρα πολύ νεολαία. Πάρα πολλούς νέους που εμφανίζονται στις ε, συνδιασκέψεις, ε, στις οθόνες κλπ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για το μέλλον να έχουμε συμμετοχή τόσο πολλών νέων. Χθε άκουσα μια πολύ ωραία συζήτηση με το, μεταξύ του Προέδρου Γιούγκερ και κάποιων νεαρών ανθρώπων από την Κροατία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Γερμανία. Κάποιοι από αυτούς όπως είπα, ε, εκφράζουν την ε, μεγάλη τους, ε, τον ενθουσιασμό τους για το Εράσμους και για άλλα προγράμματα συνεργασίας και πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτά δεν βγήκαν από το πουθενά. Είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι σαφές ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Πρέπει να υπάρχει επίγνωση αυτού του πράγματος. Κάποια άλλα σημεία είναι πάρα πολύ τεχνικά. Ίσως θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή όταν θα μιλήσουμε για την απλοποίηση και για, την, ε, για τον ενιαίο έλεγχο και για το ενιαίο κόστος. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δικαιούχος να εστιάζει περισσότερο στην υλοποίηση του έργου παρά στις διαδικασίες, στους ελέγχους, στη γραφειοκρατία κλπ. Ε, ευχαριστώ λοιπόν ε, και πάλι. Ήταν χαρά μου που βρέθηκα εδώ. Ελπίζω να έχουμε ευκαιρίες να ξανασυναντηθούμε, αλλά τουλάχιστον μπορώ να ελπίζω ότι θα φύγουμε από αυτή την αίθουσα με την ιδέα ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να αρχίσει ο τριμερής διάλογος να αρχίσει για όλα αυτά τα θέματα όσο ε, γρηγορότερα γίνεται. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ την κυρία Μιχαηλόβα επίσης. Δεν έχουμε χρόνο για συμπεράσματα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ε, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρισταμένους. Χαίρομαι ότι συμφωνούμε και με, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, των Περιφερειών και ε, Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αναφερθήκατε ε, για τον τριμερή διάλογο εμείς μπορεί να είμαστε παρατηρητές, όχι να μην συμμετάσχουμε, αλλά να είμαστε παρατηρητές, να δούμε αν μπορείτε να μας ε, δεχτείτε στον ε, τριμερή διάλογο στο μέλλον, αλλά τώρα έχουμε τις, ολοκληρώθηκε η συζήτηση μεταξύ μας και ελπίζω ότι αυτό θα προσφέρει πολλά στις περιφέρειες και στους πολίτες μας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Είναι απολύτως σαφές ότι το όραμά μας για το μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής είναι κοινή. Αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας, τις ευθύνες μας, όπως επίσης και τη σημασία που έχει να έχουν οι πολίτες τις δυνατότητες που προσφέρει η πολιτική συνοχή στο ταχύτερο δυνατό. Να είμαστε αυστηροί αλλά και ευέλικτοι και κοντά στους πολίτες. Αυτό είναι το μήνυμα που προέκυψε από τη σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε για συζήτηση. Θέλω να αναφερθώ σε δύο τεχνικά θέματα. Η συνεδρίαση Ρέτζι θα συνεχιστεί στις 12 ε, παρατέταρτο με ψηφοφορία. Λοιπόν, να, μην, να είστε εδώ. Και επίσης εμείς με τον κύριο Όσβαλτ και την κυρία Κρέλ θα κάνουμε μια ε, σύντομη ε, συνέντευξη τύπου εδώ έξω για να ενημερώσουμε τα μέσα ενημέρωσης για τη σημερινή μας συνεδρία. Λοιπόν, 12 παρατέταρτο ε, επαν, ξαναρχίζει η Επιτροπή Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Yeah.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

AUTHORWAVE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

I say welcome to all the members of Committee. Καλώς ορίζω τα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ που είστε στην ώρα σας για την ψηφοφορία. Ξέρετε ότι αλλάξαμε την ημέρησα διάταξη γιατί πολλοί συνάδελφοι είχαν διάφορες δραστηριότητες ε, λόγω των ημερίδων για τις περιφέρειες. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε την κοινή συνεδρίαση με την με τις ψηφοφορίες. <clears throat> σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού κοινών διατάξεων για τη χρήση του αποθεματικού επίδοσης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όπως ξέρετε, είχαμε αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό στις 20 Ιουνίου. Οι δύο συνσηγητές, Κρέλ και Ροε, αποφάσισαν να απορρίψουν την πρόταση. Από τις έξι επιτροπές που νομοδοτούν, οι πέντε και αυτές είναι υπέρ της απόρριψης. Έχουμε λοιπόν μόνο πέντε τροπολογίες επί των οποίων θα ψηφίσουμε. Να διευκρινίσω τη διαδικασία. Αν στηρίζετε, στηρίζετε την πρόταση απόρριψης πρέπει να καταψηφίσετε όλες τις τροπολογίες. Αν είστε υπέρ της πρότασης επιτροπής πρέπει να υπερψηφίσετε τουλάχιστον μία τροπολογία. Θέλει να πει τίποτα. Ε, Κανεί από του συνεισηγητέ Πολύ σωστά το παρουσιάσατε. Είναι ιστορική στιγμή. Για πρώτη φορά ως Ρέγγι απορρίπτουμε μία ε, νομοθετική πρόταση της Κομισιόν σε 15 χρόνια. Και το κάνουμε γιατί το παρακάνουν. Το επεκτείναμε το πρόγραμμα αυτό αλλά αυτά που προτείνονται είναι υπερβολικά. Και θα αλλάξει η κατάσταση με το νέο πι. Είναι η πρώτη φορά που η Ρέγκη στην ουσία αρνείται να εκφράσει εμπιστοσύνη προς την Κομισιόν. Ελπίζω βέβαια για να δούμε και τι θα γίνει με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε τίποτα ή να περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Ωραία, ψηφίζουμε για τις τροπολογίες. Τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά παρακαλώ. Απορρίπτεται. Τροπολογία NV1 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 ποιοι είναι υπέρ κατά παρακαλώ αποχές απορρίπτεται και τώρα τελική ψηφοφορία Ονομαστική. Άρχεται. <clears throat> Πέρας. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίπτεται. Και δούμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ψηφοφορία. Είναι η γνωμοδότησή μα. Συντάκτης ο κύριος Βόν για την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 21-27 η θέση του Κοινοβουλίου εν ώψη συμφωνίας. Κύριε Βόν, θέλετε να πείτε τίποτα. Ναι, συντόμως. Οι γνωμοδοτήσεις μας είναι σε διάφορες κατηγορίες σημασίας. Άλλε είναι σημαντικότερες από τις άλλε. Ε, αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πειράσουμε το επόμενο που Ξέρω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών περιμένει η Επιτροπή μας να υποβάλει τις προτάσεις της για να τις λάβουν υπόψη όταν θα διαπραγματευτούν το επόμενο που Είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις με τους Κιώδης και άλλους συναδέλφους και με βάση τις συζητήσεις ε, διατυπώσαμε μια σειρά από συμβαστικές πρωτολογίες άρα προς τους αδέλφους ακόμη και δεν σας ικανοποιεί πλήρως το περιεχόμενο όλων των συμβασμών παρακαλώ υπερψηφίστε αυτή τη γνωμοδότηση νομίζω πως θα ήταν τεράστιο λάθος εάν η Επιτροπή μας δεν υποβάλλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών Ξέρω ότι δεν αρέσουν όλες τις λεπτομέρειες σε όλους σας. Παρακαλώ υπερψηφίστε την τελική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος να ψηφίσουμε. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 14 πέρας εγκρίνεται Ορίστε το αποτέλεσμα. 17-14. Τροπολογία 16. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας ελέγξουμε την, την 18 ελέγχουμε άρχεται πέρας απορρίπτεται 13 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 Α, είναι ταυτόσιμη και 26, άρα έχει ήδη απορριφθεί. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Ε, 27. 27 λοιπόν έλεγα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συγγνώμη. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πιστεύω αλλά ελέγχουμε την 40 άρχεται πέρας απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πιστεύω αλλά θέλετε να ελέγξουμε Ελέγχουμε την 52. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Ωραία, ελέγχουμε την 62. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Mm. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δικό μου λάθος. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 57 ναι καταπίπτει για την εκρήθη 53 Λοιπόν, οπότε πάμε στην 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 9 υπέρ κατά Ποχές. δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή πιστεύω. 64 Α, έχει αποσυρθεί. Όπως και 65 ταυτόσιμες 66 α όχι θα την ψηφίσουμε Α, λοιπόν, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Η 64 έχει αποσυρθεί. Αλλά 65, 65 όχι. Άρα πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 λοιπόν τώρα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 67 παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε τα 67. Καλώς. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 68 και 69 που είναι ταυτόσιμες. Α, Α, καλά, α, καλά, καταπίπτουν. Οπότε, 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται αιτιολογικές σκέψεις συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή Α, θέλετε να ελέγξουμε την 3 Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε. Την πέντε. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Τι γίνεται με την έξι τώρα. Α, καταπίπτει. Οπότε πάμε στην 7. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές θέλετε να την ελέγξουμε καλά ελέγχουμε την 7 άρχεται πέρας απορρίπτεται και η 8 υπέρ παρακαλώ κατά Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Οπότε, τελική ψηφοφορία. Η οποία και άρχεται. Πέρας. Εγκρίναμε λοιπόν την απόφαση απόρριψης της πρότασης Επιτροπής. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Κλείνει τη συνεδρίαση. Θα τα πούμε στις 3. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά στις